Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος, ήρθε η ώρα να αρχίσουμε. Έχουμε και τον ε, Επίτροπο, αλλά έχουμε το πρώτο θέμα της σημερινής διαδικασίας που είναι η έγκριση αυτής. Αν δεν υπάρχει κάποια ένσταση, το σχέδιο αυτής εγκρίνεται χωρίς τροποποίηση. Ε, ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Έχουμε σε 20 γλώσσες ε, διερμηνία σήμερα και έχετε τα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο και μεταδίδεται και στο διαδίκτυο συνεδρίαση μας. Και τώρα πάμε στο τρίτο σημείο της σημερινής το οποίο είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ανδριούκαΐδης που είναι ο Επίτροπος για Υγεία και Ασφάλεια Τροφίμων στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος κύριε Επίτροπε και η ανταλλαγή απόψεων γίνεται στα πλαίσια αυτού του διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Και στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να μας πείτε τι γίνεται με την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας του 2016 και τις προτεραιότητες ε, του χαρτοφυλλοκίου σας για το έτος αυτό. Οπότε θέλουμε να μας πείτε πώς βλέπετε ε, το θέμα της αντιμετώπισης των μικροβίων και της ε, αντίστασης αυτών και ε, επίσης θα πρέπει να τι γίνεται με το θέμα της ενίσχυσης των ΜΜΕ. Θα πρέπει να ακούσουμε με ποια κριτήρια θα ρυθμιστούν κάποιες χημικές ουσίες γιατί έχουμε τις προτάσεις που θα υποβάλλεται μέχρι τον Ιούνιο και να δούμε τι θα γίνει με την υποχρεωτική ετικετοθεσία ε, των ε, επεξεργασμένων τροφίμων. Είχαμε άλλωστε και το ψήφισμά μας πρόσφατα επίσης. Πέστε μας τι θα κάνετε όσον αφορά μια νέα στρατηγική για το αλκοόλ. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ω συνήθως θα μας κάνετε μία δεκάλεπτη ε, εισήγηση. Έχετε το λόγο αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνά γρήγορα ο καιρός. Πέρασε μια ολόκληρη χρονιά από την τελευταία φορά που σας επισκέφθηκα και μιλήσαμε στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου. Πέρσι σας είπα τις προτεραιότητες που έταξα για τη διάρκεια της θητείας μου φέτος. Θέλω να περιοριστούμε σε κάποια ε, πολύ σημαντικά θέματα που μας απασχολούν. Δηλαδή, αν θέλετε, μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις μετά για όποιο θέμα νομίζετε. Για να δούμε. Με κάποια καυτά ζητήματα να δούμε τι καταφέραμε πέρσι. Πρώτα-πρώτα για την καλομεταχείριση των ζώων. Εδώ έχουμε θέμα προτεραιότητα και θέλουμε να προχωρήσουμε ταχαίω για κάποιε δράσει ούτω ώστε η σχετική στρατηγική για την καλομεταχείριση των ζώων να ολοκληρωθεί. Έχουμε επομένω πέντε δράσει από τι αρχές Ιανουαρίου. Επίση δημοσίευση των κατευθυντηρίων όσον αφορά την καλομεταχείριση των χείρων. Αυτό ήταν σημαντικό βήμα προ τα εμπρό και για το μέλλον θέλουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις δράσεις της στρατηγικής και να έχουμε μια πλατφόρμα για την οικονομική των ζώων, πρότεινα πρότειναν κάποια κράτη-μέλη, αλλά όπως έχει ζητήσει και το Κοινοβούλιο. Τώρα για το αλκοόλ, σύμφωνο μαζί σας ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε και θα πρέπει το ζήτημα αυτό να μας απασχολήσει, όπως είπαμε, και στο ψήφισμα του Απριλίου. Έχω ήδη αναπτύξει κάποια δραστηριότητα για κάποια τέτοια ε, ζητήματα με τους εμπλεκομένους αλλά και τα κράτη-μέλη και τα εθνικά κοινοβούλια και τους έχω ενθαρρύνει να αναπτύξουν δραστηριότητα όσον αφορά τον έλεγχο και έχουμε διαθέσει φέτος 1,7 εκατομμύρια ευρώ για νέες δράσεις ε, σύμφωνα με το πρόγραμμα υγείας που για να έχουμε περιορισμό τη προσβασιμότητας ε, στο αλκοόλ. Οπότε και θέλουμε να υπάρξει μια κοινή δράση η οποία θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο. Επίσης θέλουμε να υπάρξει η υλοποίηση του προγράμματος δράσης για την χρήση του αλκοόλ από τους νέους και επίσης θέλουμε να ξεκινήσουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τις γυναίκες που έχουν ε, πρόβλημα και εξάρτηση από το αλκοόλ. Τώρα, όσον αφορά την πρόληψη, εγώ έχω αποφασίσει να αναλαβώ δράση όσον αφορά την κατανάλωση των τρανς λιπαρών ουσιών. Και όπως ξέρετε αυτού του είδους τα οξέα αυξάνουν τις πιθανότητες ε, καρδιοπαθειών. Και ε, με μεγάλη μου χαρά είδαμε ότι ε, εγκρίναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια σχετική έκθεση και θα σας παρουσιάσουμε τα μέτρα μας του χρόνου βεβαίω και θέλουμε δούμε και άλλα θέματα σε σχέση με τα τρόφιμα και συνεχίσουμε την ίδια πορεία. Τέλος, όσον αφορά την οδηγία για κάποια θέματα διασυνοριακά, θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση και επίσης έχουμε μία πρωτοβουλία που θα προωθηθεί σε σχέση με τη συγκρότηση αυτών των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς. Διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών υγείας θα συνεργαστούν επομένως μέσω αυτών των διαρθρωμένων δικτύων. Ελπίζουμε να ξεκινήσει ε, η υπόθεση αυτή τέλη του 2016. Για να δούμε τώρα κάποια επίκαιρα ζητήματα. τα πότε. έχουμε κάτι το οποίο όλοι το γνωρίζετε που είναι η γλυφοσάτη. Εδώ αποκλείουν, αποκλείουν οι των επιστημόνων και αυτό γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν δεν μπορούν να καταλήξουν κάπου. Οπότε χρειάζεται η γνώμη των εμπειρογνωμόνων. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε κάποια προϊόντα προστασίας που είναι φυτικά. Και γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχει ένα σύστημα ε, επιστημονικής συμβουλής. Ε, οπότε θα πρέπει να συνεργαστούν τα θεσμικά όργανα και αυτό το σύστημα να το θωρακίσουμε όλοι μας. Ήδη έχουν ξεκινήσει επαφές μεταξύ υπηρεσιών της Επιτροπής και των κρατών μελών για το πώς θα προχωρήσουν. Οπότε γι' αυτό και θεωρώ πολύ θετικό αυτό που ψηφίσατε στην Ολομέλεια πριν από δύο εβδομάδες και επομένως θα ληφθεί αυτό υπόψη από το Σώμα των Επιτρόπων. Όσον αφορά την διαφάνεια, όπως γνωρίζετε, έχω καλέσει την βιομηχανία να δημοσιοποιήσει κάποιες μελέτες και θα έχετε προσέξει ότι, είπαμε, ότι έχουμε μια δόσμια συνέντευξη τύπου στις 4 Μαρτίου μετά από το Συμβούλιο. Και νομίζω ότι όσα είπα, ακούστηκαν από την βιομηχανία, ελπίζω θα τα λάβετε και εσείς υπόψη. Βέβαια δεν έχω αυτές τις μελέτες, οπότε δεν μπορώ να τις ε, δημοσιεύσω. Επομένω, θα πρέπει να τις ε, δημοσιεύσουν οι της βιομηχανίας. Ε, οπότε βεβαίως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα όσα εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο και η σχετική νομοθεσία. Τώρα, Να δούμε τι γίνεται με αυτές τις ενδοκρινικές ουσίες. Ε, είπαμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποια ε, επιστημονικά κριτήρια. Και πέρσι προσωπικά ασχολήθηκα με την σχετική επικοινωνία μαζί σας για το πολύπλοκο αυτό ζήτημα και οργανώσαμε μια στρογγυλή τράπεζα με ευρωβουλευτές. Κάποιοι από εσάς ήρθαν και συμμετέσχουν. Είχαμε επίσης δύο διασκέψεις για να μπορέσουμε να δουλέψουμε με συνδικής διαφάνειας. Και έτσι και θα συνεχίσουμε αξιότιμοι βουλευτές. Σας βεβαιώνω ότι δεσμεύομαι να ασχοληθώ με την προστασία της ανθρώπινης υγείας σε όσο γίνεται πιο υψηλό επίπεδο ε, ακριβώς ε, όπως ορίζει και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οπότε θα πρέπει να με βοηθήσετε κι εσείς για τις επόμενες φάσεις που θα ακολουθήσουν στο εγγύς μέλλον. Τρίτον, να δούμε τι έγινε με τον ιό Ζήκα. Έχουμε εκδώσει καθημερινές γραμμές και οδηγίες για τους ταξιδιώτες και τους επαγγελματίες του κλάδου υγείας. Κινητοποίησαμε 10 εκατομμύρια ευρώ για έρευνα, οπότε θα συνεχίσουμε ε, ε, τη συνεργασία με τον ΟΗΕ αλλά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οπότε θέλουμε να υπάρξει συντονισμός για να έχουμε όσο γίνεται λιγότερο κίνδυνο μετάδοσης στην Ευρώπη. Για να δούμε τώρα κάποιες άλλες πρωτοβουλίες ε, και αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν στους αμέσως επόμενους μήνες. Πρώτα-πρώτα η αντιμικροβιακή ε, αντοχή. Ξέρετε ότι έχουμε το πενταετές πρόγραμμα δράσης για ε, αυτή την υπόθεση, το οποίο τώρα θα ολοκληρωθεί φέτος. Οπότε θα γίνει μια εξωτερική ε, αξιολόγηση και θα σας παρουσιάσουν τα αποτελέσματα τέλη του έτους. Έχουμε επίσης μια υπουργική σύνοδο για τη μικροβιακή αντίσταση και επίσης έχουμε συμμετάσχει με τους ε, αρμόδιους υπουργούς υγείας και γεωργίας ε, σε συνεργασία με την Ολλανδική Προεδρία ούτως ώστε να υπάρξει πολιτική όθηση για το μέτωπο αυτό και τα κράτη-μέλη μας στηρίζουν. Επίσης είπαμε ότι θα πρέπει να προσέξουν τι γίνεται και με τα αντιμικροβιακά ε, από πλευρά και την ιατρική που είναι και αυτό πάρα πολύ βασικό και είπαμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτέ οι ουσίε, δηλαδή οι αντιμικροβιακέ, με μεγάλη προσοχή. Επίση, έχουμε κάποιε νομοθετικέ προτάσει για τα φάρμακα ε, τη κτηνιατρική και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία στο, στη μάχη κατά, κατά της αντίστασης ε, των μικροβίων. Επίση, έχουμε και το δικό σας κείμενο που λάβουμε υπόψη. Ε, λάβουμε μέρος στο G7 και εκεί είχαμε σημαντικές δεσμεύσεις των ε, αρχηγών κρατών και υπουργών υγείας. Επίσης η Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν συγκροτήσει αυτήν την υπερατλαντική task force και επίσης έτσι θεσπίστηκε ένα πλαίσιο συνεργασίας υπερατλαντικής ε, που θα κρατήσει πέντε χρόνια και θα συμμετάσχουμε το Σεπτέμβριο του 2016 ε, στη σχετική συνάντηση υψηλού επίπεδου του ΟΗΕ και ε, μην αμφιβάλλετε εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας και εδώ και σε διεθνέ επίπεδο. Επίσης νομίζω ότι είναι πολύ θετικό ότι σε να σας ενδιαφέρει η υπόθεση Τη αξιολόγησης της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας. Και γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να, το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα ε, εργασίας να οδηγήσει σε μια αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας και οπότε στην ανακοίνωσή μας είπαμε ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο συντονισμός, να μην ε, έχουμε επικάλυψη στις ε, αξιολογήσεις των τεχνολογιών υγείας στα διάφορα κράτη-μέλη. Και ε, με βάση την συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρούμε έναν μηχανισμό ε, συνεργασίας που να γίνει βιώσιμος από το 2020. Είπαμε επομένω ότι τώρα ζυγίζουμε την ε, συγκυρία, προσπαθούμε να επισημάνουμε τις διαφορετικές επιλογές ε, πολιτικής και θα τα συστήσουμε κατά το δεύτερο εξάμεινο του ανεστώτος έτους. Τώρα, για να δούμε κάτι άλλο. έλεγχος του καπνίσματος. Έχουμε τις προτεραιότητες για φέτος και είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, μεταφορά της ε, οδηγίας για τα προϊόντα τα καπνικά στο ε, Υπουργείο των κρατών μελών και να υπάρξει και η κατάλληλη δευτερογενής νομοθεσία και εμεί είπαμε ότι θα έχουμε κάποιες φορμοστικές πράξεις όσον αφορά την ετικετοθεσία, το, το, την συσκευασία και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Είπαμε ότι θα έχουμε ε, σύντομα έγκριση νέων ε, ε, εφαρμοστικών πράξεων και προσπαθούμε επίσης να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη ή στη μεταφορά στα αυτών των σχετικών οδηγιών. Τώρα θα πρέπει να σας επενθυμίσω ότι αργήσαμε όσον αφορά την ολοκλήρωση της έκθεσης για την αιτιοτοθεσία των αλκοολούχων ποτών και έγινε το πρώτο βήμα και αυτό είναι πολύ θετικό, είμαι έτοιμος να το συζητήσω ε, επί τη βάση του σχεδίου κειμένου που έχω εγκρίνει από την άλλη μεριά. Πολλέ φορέ έρχεστε και μου λέτε κάποια πράγματα περίεργα. Μερικοί μου λέτε ναι στην ετικετοθεσία, αλλά μόνο για ορισμένα εργολούχα ποτά. Τι σημαίνει αυτό όσον αφορά την, ε, την προστασία σε υψηλό επίπεδο τη ανθρώπινη υγεία. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, νομίζω ότι ήδη αρκετά μακρηγόρησα και τώρα περιμένω τις ε, ερωτήσεις που τυχόν έχετε. Thank you very much, Commissioner. And now we can... Ευχαριστούμε πολύ τον ε, Επίτροπο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις ε, πρώτες παρεμβάσεις και καταρχήν τους εκπροσώπους των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Κύριο Σιγκομπέλτ λοιπόν για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να θέσω ένα συμπληρωματικό ερώτημα σε ό,τι αφορά το το γνωρίζετε. Γνωρίζετε αυτή την ουσία και γνωρίζετε ότι υιοθέτησε μια ένα πολύ σαφές ε, ψήφισμα το ε, Κοινοβούλιο με πολύ συγκεκριμένες απαιτήσει έναντι της Επιτροπής. Ε, και συγκεκριμένα αναφέρει δηλαδή το ψήφισμα ότι θέλουμε η Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση νομοθετική. Και γνωρίζουμε όλοι μας ότι φτάσαμε σε ένα πολύ καλό συμβασμό μεταξύ των πολιτικών ομάδων σε ό,τι αφορά αυτό το ψηφίσμα για την, ε, για την υποστήριξη υιοθέτηση ενός ε, περιορισμένου στόχου ε, σε ό,τι αφορά το λιφόζατε. Εμεί ζητάμε από εκεί και μετά να απαγορευτούν να περιοριστούν οι χρήσεις του λιφόζατ τουλάχιστον ε, στην περίοδο πριν από τη Σωδία, γιατί ακριβώ εκείνη την περίοδο ε, εντοπίζονται και μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την υγεία. Ε, δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα έχουμε πει περαιτέρω, δηλαδή σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την μη επαγγελματική χρήση του, του γλυφοσάτ και ούτω καθεξής. Ε, επίσης θα ήθελα να σε υπενθυμίσω μια προηγούμενη ανακοίνωση από την πλευρά της Επιτροπής η οποία ανέφερε ότι δεν πρόκειται να αντιταχθεί ε, σε περίπτωση που υπάρχουν πλειοψηφίες ε, στο, στο Κοινοβούλιο. Οπότε ε, θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο θα σεβαστείτε το αποτέλεσμα αυτού του ψηφίσματος, το οποίο όπως σας είπα συγκέντρωσε μια σαφέστατη πλειοψηφία εντός του, του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Πανιό, για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Ευχαριστούμε για τις διευκρινήσεις. Ε. Θα ήθελα να ζητήσω και κάποιες ε, παραπάνω. Πρώτα απ' όλα για τα έτοιμα φαγητά και την προέλευση των, ε, προϊόντων, των ζωικών προϊόντων. Βάσει μια πρόσφατης μελέτης, Uh, uh, Έχουμε ένα πρόβλημα με τη ερμηνεία. Okay, Mr. Pagno, can you restart? Μπορείτε να ξαναρχίσετε, κύριε Παγνιό. Επίτροπε, με ακούτε τώρα. Problème technique. The technicians are trying to... Ah, static.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 ε, μιλήσω για την ετικετοθεσία στα έτοιμα ε, φαγητά σε σχέση με τα προϊόντα ζωικής ε, προέλευσης. Ξέρουμε ότι έχει αποτύχει η νομοθεσία. 54% των έτοιμων φαγητών δεν αναφέρονται καθόλου στο κρέας και 90% των σάντουιτς, παραδείγματος χάρη, δεν αναφέρουν το κρέας που έχει, την προέλευση του κρέατος που έχει χρησιμοποιηθεί. Στις 22 Μαρτίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ζητήσαμε υποχρεωτική χνηλασιμότητα. 14 Μαρτίου 2014 δόθηκε έγκριση στη Γαλλία να κάνει ένα πείραμα για τα γαλακτοκομικά και για τα ε, ζωικά προϊόντα στα έτοιμα τρόφιμα. Ε, μπορείτε να μας το επιβεβαιώσετε γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είναι οριστική η άδεια που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κανονικά χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες από τις γαλλικές αρχές και να μπορέσει να γνωμοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαντική πληροφορία. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Για τη ρύθμιση των ε, τιμών των καινοτόμων φαρμάκων, ε, ε, είπατε ότι στις 26-27 Μαΐου συνεδριάζει η G7 στο Τόκιο. Μπορείτε να μας πείτε αν προβλέπει μέτρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη σε σχέση με τον προσδιορισμό τιμών των καινοτόμων φαρμάκων. Ένα παράδειγμα να πάρουμε, παραδοσιακή θεραπεία 12 ε, εβδομάδες, ε, σοφός μπιβίρ, ένα φάρμακο για την ε, υπατήτηδα σε 5.000 στη ΣΥΠΑ, 41.000 στη ΣΥΠΑ, 40 στην ε, Ταϊλάνδη. Ε, και η Λίγα κατά του... Ο Σύνδεσμος ε, για τους καρκινοπαθείς ζητά ε, μείωση της τιμής των φαρμάκων για τον καρκίνο, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλες οι διαφορές, 100.000 το χρόνο χρειάζεται κάποιο δοκέντρωτα που είναι για τον καρκίνο του δέρματος. Είναι νομίζω σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία παρότι γνωρίζω ότι είναι εθνική αρμοδιότητα το προσδιορισμός των τιμών των φαρμάκων. Και τέλος, ε, πολύ γρήγορα, να αναφερθώ στο νομικό πλαίσιο για, τους νέο, για τα νέα μεταλλαγμένα. Μέχρι το πέρα του τρέχοντος περιμένουμε νομική αξιολόγηση σε σχέση με την, ε, το πρόγραμμα επιλογών. Μπορείτε να μας πείτε πότε θα καταθέσετε την ε, αξιολόγηση αυτή εδώ στο Κοινοβούλιο και συνέχεια στα κρατημέλη στο Σύμβουλιο. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκέρλινγκ για το ECR. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τον ε, μηχανισμό επιστημονικής, ε, επιστημονικών συμβουλών. Ε, χρειαστήκαμε πολύ χρόνο για να συγκροτήσουμε αυτό το υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμόνων που ουσιαστικά αντικατέστησαν τον Επιστημονικό Σύμβουλο του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συναποτελείται πάνω από 11 επιστήμονες, αν θυμάμαι καλά, και δεν υποβάλλει μόνο γνωμοδοτήσεις προς τον Πρόεδρο, αλλά συμβουλεύει το Σώμα των Επιτρόπων. Και σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα για την γλυφοσάτη να σας ε, ρωτήσω τι, ε, πώς, ε, προς ποια κατεύθυνση έχουν γνωμοδοτήσει, διότι είναι αντικρουόμενες οι επιστημονικές πληροφορίες που έχουμε και είναι ενδιαφέρον να ξέρουμε τι γίνεται με τις διαβουλεύσεις σε αυτή την ομάδα υψηλού επίπεδου και γενικότερα διότι καλούμεθα να αποφανθούμε παρότι υπάρχουν δύο διαφορετικές μέθοδοι δοκιμής και δύο διαφορετικές επιστημονικές απόψεις. Μήπως θα έπρεπε να τους καλέσουμε και να λάβουμε συμβουλές ή τουλάχιστον όχι σε εμά άμεσα, αλλά να λάβετε εσεί συμβουλέ σε σχέση με το πώ πρέπει να κινηθείτε. Και στη δεύτερη συνεδρία από ό,τι κατάλαβα, στα πρακτικά φέρετε ε, δηλαδή ύπουλα στα διάφορα, ε, ότι μιλάγανε για την επιστημονική αποτίμηση της γλυφοσάτης ε, και είπαν ότι θέλουν να αποφύγουν οποιαδήποτε επικάλυψη, αυτό ήταν ξεκάθαρο. Όμως θέλω να ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούσατε εσείς να χρησιμοποιήσετε αυτή τη νέα δομή. Είναι καινούργια και το ξέρω. Πιστεύω όμως ότι είναι ιδανική ευκαιρία για να χρησιμοποιήσουμε αυτό το νέο μηχανισμό, αυτή τη νέα ομάδα, ούτω ώστε να έχουμε πληροφορίες στη διάθεσή μας. Όχι μόνο εμείς, αλλά και εσείς και το Σώμα των Επιτρόπων. Θα χρησιμοποιείτε λοιπόν γι' αυτό το λόγο αυτήν την ε, ομάδα υψηλού επίπεδου ε, και πώς διαμορφώνεται το μέλλον κατά τη γνώμη σας αυτού του νέου μηχανισμού επιστημονικών συμβουλών. Σας ευχαριστούμε από τους φιλελεύθερους. Η κυρία Χρυσέ, ε, ευχαριστώ πρόεδρε, επίτροπε. Ε, πάντοτε χαιρόμαστε όταν σας βλέπουμε εδώ στην Επιτροπή μας, διότι μας διαφωτίζετε για ζητήματα που μας απασχολούν και ε, σίγουρα δεν θα είμαι η μόνη, συγχωρέστε μας. Θέλω και εγώ να ε, μιλήσω για το μάτι κυκλώνα, για την κλειφωσάτη. Ε, αρχίσατε με αυτό το ζήτημα, με αυτή την καυτή πατάτα, όπως λέμε στα αγγλικά. Ε, συζητείτε το ζήτημα διυπηρεσιακά στο Σώμα των Επιτρόπων και θα λάβετε υπόψη τη ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Την περασμένη Παρασκευή... Ε, είδαμε δημοσίευματα τύπου για μια υποτιθέμενη απόφαση τη ομάδα εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια νέα πρόταση που θα καταδεχθεί στα κράτη-μέλη για την κρίσιμη συνεδρίαση τη 17η Μαου, δηλαδή η έγκριση, αδειοδότηση για 10 χρόνια, όχι 5, 7, 10 χρόνια, δεκαετή αδειοδότηση. Η Επιτροπή δεν μιλάω για εσά γιατί ξέρω ότι Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε εσά και το σώμα των επιτροπών. Εντάξει να μην ακούνε το κοινοβούλιο, να μην ακούνε του εμπειρογνώμονε, να μην ακούνε τι μη καπαόμικρον, αλλά να μην βλέπουν και τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Σε πάρα πολλά κράτη-μέλη, η Γερμανία, η Πολωνία, η Δανία και σύντομα και το Βέλγιο και η Γαλλία έχουν τέτοιε πρακτικέ κατά ε, τη χρήση αυτού του ζυζανιοκτώνου. Οπότε όταν ε, μας λέτε ότι θα ληφθεί υπόψη αυτό που υπάρχει ω προ τη συμβαστική του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σε σιγουρευτείτε ότι θα γίνει και κάτι άλλο για τα καπνό και τα προϊόντα το Είμαστε στην κρίσιμη περίοδο της μεταφορά στην Εθνική Νομοθεσία και υπογράψαμε το Δεκέμβριο του 2013. εσεί ήσασταν στο Συμβούλιο τότε. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσω για το ουδέτερο πακέτο στα ε, υπάρχουν τα κράτη-μέλη που έχουν εφαρμόσει ήδη αυτό το στην νομοθεσία για την ε, ουδέτερη ετικετοθεσία στο πακέτο. Εσείς ε, τι πιστεύετε για αυτά τα ε, ε, γενώσιμα, πούμε, πακέτα τσιγάρων και για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Επίση, θα ήθελα να τοποθετηθείτε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν σοβαρέ διαστάσει απόψεων για αυτά τα ζητήματα και εξ αρχή θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ό,τι μπορούσε για να εμποδίσει την ανάπτυξη αυτή τη αγορά ε, γιατί ε, το χαρακτήρισε σχεδόν ω φάρμακο το ηλεκτρονικό τσιγάρο και για τα μέσα Μαΐου είχατε υποσχεθεί κάτι. Δεν περιμένω πολλά πράγματα διότι εξ αρχή ε, προσδώσατε ιδιαίτερη σημασία στην διάσταση του κινδύνου. Λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, μετά τι αξιολογήσει σε επιστημονικέ, όχι από τον καθηγητή Βόλσεμπεργκ, όχι από τον καθηγητή West ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Βέλιο και σε πάρα πολλέ χώρε, ε, βλέπουμε ε, γνωμοδοτή που λένε φυσικά ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο θα πρέπει να απαγορεύεται για του νέου θα πρέπει να είναι προσβάσιμο για όσοι το χρειάζονται, σημαίνει απλώ και μόνο αρχή τη πρόληψη. Αυτό το λάβατε υπόψη σα, στην αξιολόγησή σα Ευχαριστούμε. Μπόιλαν Γκουαρτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε ε, τον Επίτροπο και τον ε, ευχαριστώ ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ε, πολιτική για τα Ε, και θα ήθελα να λάβω και κάποιες περισσότερες πληροφορίες με βάση την επικείμενη στρατηγική για τα Ε, Εκεί αναφέρεται δηλαδή το κενό που υπάρχει σε ό,τι αφορά τα το δίκαιο το κατά πόσο καλύπτονται από την νομοθεσία για τα τρόφιμα. Αυτό λοιπόν το νομοθετικό κενό μα έχει οδηγήσει σε αυτήν την ε, ε, περίεργη κατάσταση του να έχουμε περισσότερε πληροφορίε διαθέσιμε για το καταναλωτή όταν αγοράζει ένα μπουκάλι γάλα από ότι όταν αγοράζει ένα μπουκάλι κρασί. Ε, και νομίζω πως το ότι αποχώρησαν οι NGOs, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις από την σχετική συνεδρίαση των εμπλεκομένων φορέων λέει πολλά για το πού βρισκόμαστε και νομίζω πως ε, κύριε Επίτροπε, ε, ε, εσείς καθώς είστε εκείνο ο οποίο προβαίνει σε συζητήσει με τους Υπουργού Υγεία για τα ζητήματα των πνευματοδών, να σας ρωτήσω, θεωρείτε πως προβλέπετε ένα τέτοιο σχέδιο δράση σε ό,τι αφορά το πώ μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερο αντίκτυπο των Ε, Η υπάρχει και η αξίωση μέσα στη σχετική έκθεση σε ό,τι αφορά την ετικοτοθεσία των ίνοπνευματοδών και γνωρίζουμε πως αυτό το ζήτημα είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τους καταναλωτές, οπότε θα θέλαμε ε, να μας ε, πει η Επιτροπή να μας δώσει μια συγκεκριμένη ημερομηνία ως προς το πότε να αναμείνουμε αυτή την έκθεση για την ετικοτοθεσία. Επίσης αναφερθήκατε σύντομα σε ένα σχέδιο δράσης σε ό,τι αφορά τη χρήση ινοπνευματοδών από τους νέους. Λαμβανομένο υπόψη του γεγονότος ότι τα ε, ορισμένα κράτη-μέλη έχουν προσπαθήσει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα του, της υπερβολικής λήψης πνευματοδών, ε, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη χρήση τους από νέους. Θα ήθελα να μας πει η Επιτροπή ποια είναι η άποψή τους σε σχέση με ε, τις προσπάθειες που κάνουν συγκεκριμένα κράτη-μέλη, οι οποίες είναι πραγματικά υψηλότερες του μέσου σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της ε, ε χρήσης πνευματοδών. καθώς βλέπουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν οδηγηθεί ενώπιον ε, του δικαστηρίου ε, της Ευρωπαϊκής, μόνο, ε, μόνο και μόνο επειδή προσπάθησαν να προστατεύσουν καλύτερα τους τους. Ευχαριστούμε για τους πράσινους κύριε ε, Ευχαριστώ. Ε, εμείς έχουμε τονίσει το ζήτημα των ουσιών ενδοκρινικής διαταραχής από την αρχή της εντολής σας, αλλά ε, δυστυχώς η Επιτροπή ακόμα δεν έχει οθετήσει επιστημονικά κριτήρια, ε, ε, όπως είχε προς το 2013. Υπήρξε μια απόφαση ε, το 2013 μετά από πιέσεις του κλάδου για να υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια. Όμως είναι ε, παράλογο το να υπάρχει μια αξιολόγηση αντικτύπου για ένα επιστημονικό ζήτημα και το δικαστήριο είπε συγκεκριμένα ότι δεν ε, χρειάζεται αξιολόγηση αντικτύπου. Παρ' όλα αυτά η Επιτροπή αποφάσισε να προβεί σε, μια, σε αυτή την αξιολόγηση αντικτύπου. Δηλαδή είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να αγνοήσει ακόμα και την απόφαση του δικαστηρίου εάν αυτό της επιτρέψει να βοηθήσει ε, την, τον κλάδο των φυτοφαρμάκων ε, προκειμένου να μην κλείσει το θέμα όπως είχε αρχικά προβλεφθεί το 2009. Ένα ε, σημαντικό ζήτημα ε, για μας είναι στο μέλλον και η ισχύς. Για παράδειγμα, εκπρόσωποι ε, και από τις δύο πλευρές ε, τη συζήτηση αυτή ε, για τι ουσίες τη ενδιοκρινικής διαταραχή, έφτασαν σε μια πρώτη συμφωνία στο Βερολίνο. Ε, δηλαδή θεώρησαν ότι δεν χρειάζεται να, να λάβουμε υπόψη μας το ζήτημα τη ισχύω για να ορίσουμε τον endocrine disruptor και νομίζω πως μπορείτε τώρα να αποκαταστήσετε την εμπιστοσύνη της Επιτροπής εάν τουλάχιστον δεν συμπεριλάβετε σε αυτή την αξιολόγηση αντικτύπου σας το ζήτημα της ισχύω σε ό,τι αφορά τον ορισμό των ουσιών αυτών. Μπορείτε λοιπόν να μου υποσχεθείτε ότι αυτός ο παράγοντας της ισχύω δεν θα ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο του ορισμού των ουσιών ενδοκρινικής διαταραχής. Εάν όμως το κάνετε, αν δηλαδή ε, τι συμπεριλάβετε, την πότε στην ισχύ, ε, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ασκήσουμε βέτο, γιατί για μας θα έχει λήξει εκεί το θέμα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, κύριος για το EFTD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε που είπατε για το πόσο έχει δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ε, καταπολεμήσει την ανθεκτικότητα των μικροβιολόγων των ε, αντιβιωτικών που τη χρήση με τελευταία ανταγωνική ακριβώ, όπω έχει πολλέ φορέ επαναληφθεί όσον αφορά τι επαφέ μα με του γιατρού και με του κτηνιάτρου. Θα, ε, πιο καλό είναι να ανοίξει μια αγορά παρά να κλείσει. Οπότε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να μην υπάρχουν καταχρήσει ε, από μονοπόλια της φαρμακοβιομηχανίας και, ε, ε, και να κλείσουν οι ανεξάρτητοι φορείς. Οπότε τέτοια πολιτική πρέπει να κάνουμε και εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποιο ευρωπαϊκό επιμελητήριο για να ελέγξει τα πράγματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει και έρευνα όσον αφορά τα φυσικά αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται στην ιατρική και πέραν της κτηνιατρικής. Έχουμε επίσης και την έκθεση που έγινε πέρσι ε, όσον αφορά την ε, ασφάλεια στα θέματα υγείας και φαρμάκων. Οπότε θα πρέπει να μας πείτε εσείς ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα κάνετε. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε, Επίτροπη, λέει η κυρία Αντωνάνου. Αναφερθήκαμε ήδη σε διάφορα ζητήματα, αλλά όχι αρκετά κατά τη γνώμη μου. Το αλκοόλ και η ευρωπαϊκή στρατηγική ε, υπέρ της οποίας έχουν αποφαθεί διάφοροι βουλευτές. Ε, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι είναι σοβαρότατο το πρόβλημα, κυρίως για τους νεότερους και το θέμα δεν είναι ε, το πόσες θερμίδες έχει το ποτό, αλλά η ποσότητα που καταναλώνεται και ισχυρή κατανάλωση σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, αυτή τη συνήθεια των νέων. Ε, σε αυτό το τομέα Υπάρχει επίσης λόγω του λαθρεμπορίου ε, μεγάλος πληθωρισμός ε, και μπορούμε να πούμε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ε, να καταπολεμήσουμε την πώληση του νοθευμένου αλκοόλ και θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τη στρατηγική για το αλκοόλ να εξετάσει τα δύο εξή ζητήματα. Ε, στόχευση των νέων, να εξετάσει ποιοι εθνικοί μηχανισμοί ήταν αποτελεσματικοί μέχρι στιγμής και ως εκ τούτου ποιες συστάσεις μπορεί επί τη βάση αυτών να ε, καταθέσει. Δεύτερον, ε, τιμή, μία αξιολόγηση του κινδύνου της ενδεχόμενης αύξησης ε, της τιμής του αλκοόλ, κυρίως για τα ενεπνευματόδη και τα Υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Ε, Ποιε επιπτώσει πιστεύετε ότι θα έχει σε σχέση με την ειχνηλασιμότητα, όπω μα είπε και ο κύριο Παρνιό, ε, για τα προϊόντα ζωική προέλευση. Ε, υπάρχει τελετουργική σφαγή των ε, ζώνων σε ορισμένους κουλτούρες χωρίς ε, πρώτα να ε, αναισθητοποιείται το ζώο, ε, θα ήθελα να πάρει στα σοβαρά επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, το ζήτημα και να ακολουθήσει μια προσέγγιση δύο στάδιων. Πρώτον, να καταργηθούν αυτές οι τελετουργικές θυσίες και δεύτερον, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ξέρουν ακριβώ εάν σφαγιάστηκε ναι ή όχι το ζώο με αυτόν τον τρόπο και να αναφέρεται αυτό σε συγκεκριμένη ετικέτα. Εάν θα πρέπει να θεσπίσουμε Περιορισμού σε αυτό το τομέα. Αυτό θα ήθελα να ξέρω για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Κατόπιν, διαχείριση των επιδημιών. Όσο περισσότερο κυκλοφορούμε και όσο μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση υπάρχει, τόσο εντείνεται το φαινόμενο των επιδημιών. Είναι τόσο ισχυρέ οι μεταναστευτικέ ροέ και ε, δεν, ε, τα κέντρα υποδοχή, τα κέντρα κράτηση, τα κλειστά αυτά κέντρα δεν ε, παρκούν για να συγκρατήσουμε αυτέ τι επιδημίε. Επίση, χρειάζεται δράση για την πρόληψη, διότι είναι ουσιαστικό ο κίνδυνο. οι κομιστές είναι ε, πολλαπλοί και ε, δεν, ε, αντί να υποδεχόμαστε τη μιζέρια από όλο τον κόσμο, να αποφύγουμε τις επιδημίες για τους πολίτες μας και θέλω να ξέρω τις προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τον πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Θα ακούσουμε τώρα τον Ευρωπαϊκό για τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Επίτροπος. Ας ε, ξεκινήσουμε από την πρώτη ερώτηση του κυρίου Ιβομπέλη για την γλυφοσάτη. Βεβαίω. Και εγώ ε, θεωρούσα ότι είναι κάτι πάρα πολύ θετικό το ψήφισμά σας για την γλυφοσάτη και επίσης για τις συμβαστικές τροπολογίες και προτάσεις για την ε, περισσότερη ευελιξία. Βεβαίω και όλα αυτά πρέπει να συζητούνται. Ακριβώς σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα με τα κράτη-μέλη και σε επίπεδο της ε, Επιτροπής σας ε, βλέπω πώς ε, ψάχνονται, πώς θα έχουμε ευρύτερους συμβασμούς και συνένεση. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να συστρατεύσουμε όσο γίνεται πιο μεγάλη πλειοψηφία κρατών μελών για την τελική απόφαση. Επίσης, θα ενημερώσω το Σώμα των Επιτρόπων. Ακόμα πάντως δεν υπάρχει επίσημη απόφαση. Γίνονται απλώς επαφές μεταξύ των επιμέρους υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε να λάβουμε υπόψη όλα τα δεδομένα και έτσι να σχηματιστεί αυτή η επιθυμητή ευρεία συνένεση. Θα δούμε πώς τελικά θα έχει κάποια λογική αυτή η απόφαση και θα αγκαλιάσει από παντού αυτό το περίπλοκο θέμα. Δεύτερη ερώτηση. Κύριος Παρνιό, μας είπε για την ότι θέλει περισσότερη ενημέρωση. Είναι θέμα φυσικά ενημέρωσης του καταναλωτή όσον αφορά τα είδη διατροφής και αυτό δεν ισχύει μόνο για το βόλιο, αλλά ισχύει για το χείριο, ε, για τα πουλερικά, για το πρόβιο και είπαμε θέλουμε την πιο βιώσιμη λύση σε, για όλες τις κατηγορίες ειδών διατροφής και αυτό να γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν τα κρατημέλη να έχουν και δικά τους μέτρα, όπως είπατε και εσείς. Κάποια κρατημέλη είπαν ότι θέλουν να έχουν υποπιλωτική μορφή την υποχρεωτική ετικετοθεσία. Αυτό με ενδιαφέρει πολύ να δω πού θα καταλήξει ως πείραμα. Η Γαλλία ήδη έχει παρουσιάσει τις προτάσεις της, ε, η Ιταλία επίσης και εμείς είμαστε σε θέση αναμονής μια που ορίζονται στον κανονισμό οι σχετικοί κανόνες Οπότε, να δούμε, θα υπάρχει αναλογικότητα. Από την άλλη μεριά υπάρχει νομική υποχρέωση. Και όπως είπα θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη τέτοιων πειραμάτων. Βέβαια έχουμε και τις ε, λεπτομέρειες της εφαρμογής του κανονισμού, οι οποίες ακόμα δεν έχουν καθοριστεί. Όμως οι συνεργάτες μου πάνω σε αυτό ε, δουλεύουν και ελπίζουμε μέχρι τέλους του έτους θα έχουμε το νομικό πλαίσιο. Επίσης είπαμε για κάποιο είδους καινοτόμα φάρμακα για την πρόσβαση ε, στις ε, θεραπευτικές αγωγές, πώς θα μπορέσουμε, είναι το ερώτημα, να διευκολύνουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πρώτα-πρώτα την ομάδα εμπειρογνωμόνων. Συνέταξαν αυτοί μια έκθεση όσον αφορά έναν ε, μηχανισμό τιμολογική πολιτικής για όλα τα κράτη-μέλη και υπάρχει και κάποιο πρόγραμμα το οποίο ε, έχει ε, εκούσια μορφή για τα καινοτόμα φάρμακα. Είναι λοιπόν εκούσια και η συμμετοχή και θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό πως ολένα και οι περισσότερες χώρες προσχωρούν σε αυτό το πρόγραμμα. Και νομίζουμε ότι με τα προγράμματα τα οποία έχουμε ξεκινήσει θεωρούμε ότι είναι πιο εύκολο τώρα να εγκριθούν ε, όσο γίνεται περισσότερα φάρμακα. 18 Απριλίου είχαμε το άτυπο συμβούλιο και εκεί έγινε μια συζήτηση όσον αφορά την διαφάνεια στην τιμολογική πολιτική και είπαμε ότι θα πρέπει να αυξηθεί ε, επ' αυτού η συνεργασία των κρατών μελών και όσον αφορά την επιστροφή των ιατρικών εξόδων. Ενδιαφέρονται τα κράτη-μέλη, όλο ένα και περισσότερο. Έχουμε επίσης και την συνεργασία των χωρών Μπενελούξ από αυτό. Ο Γάλλος Υπουργός πρότεινε επίσης συνεργασία και επαφές σε επίπεδο G7 να υπάρξει ε, επεξεργασία του θέματος για τα κοινοτόμα φάρμακα. Οπότε βλέπετε πόσο σημαντική ήταν αυτή η έκθεση της ε, ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα θέματα τιμής των φαρμάκων στις 28 χώρες μέλη. Δεν θα έρθουν τα μελη να συνεργαστούν από αυτού γιατί πολλές φορές έχουμε παράλογα μεγάλη διαφορά τιμής από χώρα σε χώρα. τα φυτά τώρα και τις, ε, τους νέους τρόπους παπλασιασμού, τις νέες τεχνικές και είπαμε ότι έχουμε κάποιους νέους σπόρους που έχουν ιδιαίτερα μεγάλη ανθεκτικότητα. Άρα ε, εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ε, λιγότερη χρήση φυτοφαρμάκων. Έχουμε προβεί στην νομική ανάλυση που επιβάλλεται πάντα στα πλαίσια της ε, κοινωτικής νομοθεσίας για τις ε, μεταλλαγμένες ουσίες. Και θα υποβάλουν προτάσεις κατά τη διάρκεια του ενεστώτος έτους, γιατί είναι βέβαια απαραίτητο να ξεκαταστεί το τοπίο. Θα πρέπει να υπάρξει βιώσιμη καινοτομία για να πετύχουμε τους στόχους της βιωσιμότητας. Άρα θα πρέπει να υπάρξει προβληματισμός και μελέτη του προβλήματος αυτού. Επόμενη ερώτηση. Συμφωνώ μαζί σας. Θα πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη προς την επιστήμη όσον αφορά την αξιοποίηση των επιστημονικών στοιχείων. Υπάρχουν όντως αποκλήσεις μεταξύ των επιστημόνων αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε γιατί πολύ σπάνια ε, είναι αδιάστατα στοιχεία των επιστημονικών μελετών. Και έχουμε έναν μηχανισμό επιστημονικής παροχής συμβουλών για να δούμε πώς αυτός ο μηχανισμός θα αποδώσει και θα έχουμε περισσότερη διατροφική ασφάλεια. Θα δούμε στις λεπτομέρειες επομένω το πρόβλημα, να δούμε πώς αυτό το μηχανισμό θα τον αξιοποιήσουμε. Και πώς οι επιστήμονες που έχουμε θα μπορέσουν όλους τους και ενδιαφερομένους να τους ενημερώνουν. Άλλη ερώτηση. Η κυρία νομίζω το είπε. για την εφαρμογή και μεταβάση του ιστορικό δίκαιο. είπαμε ότι 8 κράτη-μέλη έχουν ε, το κάνει στο Βέλγιο, Εστονία, Λιθωνία, εν μέρη έχουν μεταφέρει, Γερμανία, Ιταλία, ε, Σλοβακία, Μάλτα έχουν μεταφέρει πλήρω ε, το κοινωτικό δίκαιο, άλλε χώρε μέλη, πιο προχωρημένη φάση και συζητείται το νομοθέτημα στα εθνικά κοινοβούλια, οπότε θεωρούμε ότι ε, τα περισσότερα κρατημέλη έγκαιρα θα έχουν εφαρμόσει και την νομοθεσία. Και εμείς βέβαια ενθαρρύνουμε τα κρατημένη προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα στον αφορά ε, την συσκευασία και σε σχέση με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα πολλά κρατημέλη έχουν ξεκινήσει την ε, εφαρμογή των όσων έχουμε προτείνει και άρα αυτό το βλέπουμε πολύ θετικά. Αλλά ειδικά για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, όπως γνωρίζετε, εξαρτάται από τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν και να νομοθετήσουν σχετικά. Πρέπει να υπάρχει συλλογή των δεδομένων και πληροφοριών από τους ε, ειδικού και από τις σχετικές ε, υπηρεσίες, οπότε να υπάρξει και η απαραίτητη νομοθεσία. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να διέπεται ε, από όσο γίνεται πιο αυστηρή νομοθεσία το ηλεκτρονικό τσιγάρο γιατί είναι επικίνδυνο για την δημόσια υγεία. Άλλη ερώτηση. Hm? Uh, uh, uh, about alcohol use. Α, ρωτήσατε ε, για την κατανάλωση νοπνεύματος, ε, για την τιμή ε, του υνοπνεύματος. Βεβαίω και θα πρέπει να συνεργαστούμε, να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και είπαμε θα υπάρξει κοινή δράση με όλα τα κράτη-μέλη βοηθούμε τα κρατη να εφαρμόσουν το πρόγραμμα δράσης. Τώρα όσον την ελάχιστη τιμή μονάδας, όπως ρωτήσατε, θέλουμε να υπάρχει αναλογικότητα και άπαξ και υπάρχει αναλογικότητα είναι στη διακριτική των κρατών μελών. Θέλουμε να παρακολουθήσουμε, να δούμε τι θα κάνουν τα κράτη-μέλη. Γιατί έχουμε και την απόφαση που εκκρεμεί στο Σκοτσέζικο Δικαστήριο. Οπότε θα ολοκληρώσουμε την οδηγία για την αιτιοδοσία. Θα συνεργαστούν σχετικά οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα δούμε μάλλον στο τρίτο τρίμηνο του 2016 τι απόφαση θα ληφθεί από πλευρά της Επιτροπής για την Ετικετοθεσία των Αλκοολούχων Ποτών. Επίσης όσον αφορά την χρήση και κατάχρηση του αλκοόλ, τα κράτη-μέλη έχουν υποχρέωση να έχουν επιβάλει κάποια μέτρα χρηματοδοτική πολιτική, φορολογική πολιτική, τιμολογική πολιτική όσον αφορά την πρόσβαση και τι ε, διαφημίσει. Όλα αυτά είναι μέσα πολιτική, τα οποία όμω είναι εθνική αρμοδιότητα. Και είπαμε τώρα για το θέμα της διασυνορικής ε, διαφήμισης. Αυτό τώρα το επεξεργαζόμαστε, το συζητούμε και θα καλυφθεί στα πλαίσια της ε, οδηγίας για τα οπτικοακουστικά. Πάντως, ενθαρρύνουμε τα κρατημέλη να χρησιμοποιήσουν ε, τα εργαλεία της αγοράς για να συγκρατήσουν την κατανάλωση ε, αλκοολούχων ποτών, ώστε να περιοριστεί η κατάχρηση και οι βλαβερές συνέπειες. Για άλλη μια φορά σας επαναλαμβάνω τα με έχουν κάποια δραστηριότητα και γνωρίζουν ποια μέσα πολιτική είναι πιο αποτελεσματικά. Γιατί η τιμολογική πολιτική είναι ένα εργαλείο πολύ αποτελεσματικό, αλλά είναι στην κρατική ευκαιρία των κρατών μελών. Είχαμε τώρα άλλη μια ερώτηση από την κυρία Όκεν για την γλυφοσάτη και την μελέτη επιπτώσεων. Α, όχι, όχι, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Για τους ενδοκρινικού διαταράκτε, μας είπατε και τη σχετική μελέτη επιπτώσεων. σα ευχαριστώ πάλι και για αυτή την ερώτηση. Εμείς έχουμε λάβει υπόψη την δικαστική απόφαση. Αλλά δεν θεωρούμε ότι εμείς ενεργούμε ενάντια σε αυτή την απόφαση. Είναι δουλειά μας να κάνουμε αυτή τη μελέτη επιπτώσεων και μας βοηθά. Ούτως ώστε να λάβουμε κάποια απόφαση όσο γίνεται πιο πλήρη. Βέβαια. Για τα, κριτήρια που θα λάβουμε υπόψη θα σεβαστούμε την απόφαση. αλλά δεν νομίζω ότι η πρωτοβουλία μας έρχεται σε σύγκρουση με την απόφαση. Θέλουμε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία για το περίπλοκο αυτό θέμα, ακριβώ όπως και για την ισχύ των διαταρακτών. Έχουμε τους εμπειρογνώμες που εξεργάζονται το θέμα και συνεργαζόμαστε με τοξικολόγους και στις 11 ε, Απριλίου τοξικολόγοι, ενδοκρινολόγοι ε, κάτσαν γύρω από ένα τραπέζι σε ένα συμπόσιο για να ληφθεί μια ε, απόφαση. με είμαστε όργανο νομοθετικό. Δεν έχουμε αρμοδιότητα έκδοσης κάποιας επιστημονικής γνωμοδότησης. Οπότε λαμβάνουμε υπόψη τόσο λένε οι ενδοκρινολόγοι, όσο λένε οι τοξικολόγοι. Ε, πάντως δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε ποια θα είναι τα κριτήρια που πρέπει να προτιμηθούν έναντι άλλων κριτηρίων. Ακόμα για την ισχύ αυτών των ουσιών δεν έχουμε λάβει ακόμη απόφαση. αναμένουμε την τελική έκθεση των ειδικών. για την αντιμικροβιακή ανθεκτικότητα και αυτό που είπε και ο κ. Πεντιτσίνη. Και πώς θα βοηθήσουμε τη βιομηχανία να παραγάγει νέα αντιβιωτικά. Όπως γνωρίζετε, έχουμε την σχετική πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα. Βοηθούμε, ενθαρρύνουμε την έρευνα για τα νέα αντιβιωτικά. Τώρα όσον αφορά τις δυνατότητες εποπτείας της χρήσης των αντιβιωτικών ε, στην ιατρική, μέσα το φθινόπωρο πρόκειται να ε, ε, παρουσιάσουμε κάποιες καθητήρες γραμμές για την ε, ορθή χρήση των αντιβιωτικών πλευράς της ιατρικής. Θέλουμε να υπάρξει ένα καινούριο επιχειρησιακό μοντέλο, επιχειρηματικό μάλλον μοντέλο, όσον αφορά την παραγωγή των νέων αυτών αντιβιωτικών. Γιατί από πλευρά βιομηχανία δεν υπάρχει τόσο έντονο ενδιαφέρον για παραγωγή νέων αντιβιωτικών. Πάντως εμείς συνεχίζουμε τις επαφές με όλους τους Και πάλι ρωτήσατε για την στρατηγική μας όσον αφορά τα αλκοολούχα ποτά. Συμφωνώ, συμφωνώ. Θα πρέπει να μελετήσουμε στα 28 κράτη-μέλη ποια είναι η τιμολογική πολιτική, αλλά και εμείς αναζητούμε μια κοινή στρατηγική όσον αφορά τη διαχείριση των παραγόντων του κινδύνου για, από το κάπνισμα, τα τρανς, ε, λιπαρά κλπ. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα βασικά μέσα πολιτικής για την μείωση των παραγόντων κινδύνων είναι θέματα εθνικής αρμοδιότητας, τα οποία μέλη θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η φορολογία, μέσα της πρόσβασης στην αγορά, η νομοθεσία για τη διαφήμιση, ότι όλα αυτά τα μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν δεόντως ούτω ώστε να συγκρατηθεί ο κίνδυνο και από το αλκοόλ από τα ε, ποτά. Και ακριβώ συμφωνώ με σας ότι είναι θέμα του να στοχεύει η τιμολογική πολιτική τους νέους. Επίσης για την τελετουργική σφαγή έχουμε μια έκθεση και λέμε ότι έχουμε κάποιες παρεκκλήσεις ανά μέλος. Δεν θα πρέπει να γίνεται κατάχρηση αυτών. Ο έλεγχος της φαγής είναι εθνική αρμοδιότητα. Το θέμα θα συζητηθεί και στο μέλλον στα πλαίσια της πλατφόρμας για την καλομεταχείριση των ζώων. Γι' αυτό και εμείς άλλωστε ε, θέλουμε να προσεχθεί το θέμα. Για τις επιδημίες Έχουμε έναν πάγιο μηχανισμό ελέγχου όλων των πληροφοριών για τους κομιστές και πρόγραμμα πάντως στην εκδόση οδηγιών για το πώς να γίνονται οι απολυμάνσεις και επομένως με κάθε μέσο να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τους κομιστές ή τους φορείς τέλος πάντων. Υπάρχει θέμα και πρόβλημα για το ΖΙΚΑ γιατί έρχεται το καλοκαίρι, οπότε και γι' αυτό και επαγρυπνούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον ε, Επίτροπο. Έχουμε τώρα ένα κατάλογο 21 ομιλητών, οπότε θα ήθελα να ζητήσω από όλους σας να είσαι όσο το δυνατόν ε, πιο σύντομη. Η κυρία Γκροστέτ παίρνει πρώτο λόγο. Ευχαριστούμε, Επίτροπε, που ήρθατε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σα μιλήσω για την νομοθεσία για τα κτηνιατρικά φάρμακα, διότι ακούγονται εξαιρετικά ανησυχητικά πράγματα από πλευρά Συμβουλίου. Δεν βιάζεται το Συμβούλιο. Κατά πάσα πιθανότητα θα περιμένουν το τέλο του 2016 μέχρι να καταλήξουν σε συμφωνία και άρα ο τριμερή θα αρχίσει το 2017. Παρακαλούμε λοιπόν να ασκήσετε πίεση στο Συμβούλιο, διότι μιλάμε για την ε, αντιμικροβιακή αντίσταση και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω για την αποτίμηση της ε, προσθέμενης αξίας ε, των φαρμάκων HTA, αλλά κυρίως για τα καινοτόμα φάρμακα και τα εξατομικευμένα φάρμακα. Θέλουμε να υπάρξει ταχύτατη πρόσβαση για τους ασθενείς σε αυτά τα φάρμακα. Αυτό τι σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ενδεχομένως πιο ρεαλιστικά μοντέλα για την αδειοδότηση και τη θέση σε εμπορία, χωρίς φυσικά να θέσουμε κινδύνο για την υγεία των ασθενών. Στη Γαλλία έχουμε σχετική εμπειρία για την διαδικασία προσωρινής ε, αδειοδότησης. Ξέρουμε ότι ο Ευρωπαϊκός ε, Οργανισμός Φαρμάκων πειραματίζεται τώρα με εξελικτικές ε, δραστικές ουσίε. Επίση, κάτι άλλο που με ανησυχεί, δύο κατηγορίε ειδική διατροφή ε, για τα παιδιά σε χαμηλή ηλικία και για τους αθλητέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είχε υποσχεθεί δύο εκθέσεις ε, για τον Ιούλιο του 2015. Θα ολοκληρώσω, είναι σημαντικό για τους αθλητές και την ειδική διατροφή. Δεν υπάρχει αυτή η έκθεση, ενώ το ενισχύει κανονιστικό πλαίσιο θα εκπνεύσει τον Ιούλιο του 2016. Τι θα συμβεί λοιπόν και για τα παιδιά σε χαμηλή ηλικία, δημοσιεύθηκε η έκθεση πρόσφατα και προτείνει εγκατάλειψη του ε, ειδικού ρυθμιστικού ε, πλαισίου. Μα αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Δεν θα υπάρχει δηλαδή ειδική νομοθεσία για τα τρόφιμα για τα παιδιά σε χαμηλή ηλικία. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο και περιμένουμε λοιπόν να δράσετε σε αυτό το τομέα. Ο κύριος Λαβία, σας παρακαλώ να είσαστε σύντομοι συνάδελφοι. Ο κύριος Πότς. Αξιότιμη κυρία Επίτροπε. είδα ότι λάβατε πάρα πάρα πολλές ε, ερωτήσεις σε σχέση με την Κλειφόζάτη Αλλά ε, δυστυχώς θα πρέπει και εγώ από την πλευρά να αναφερθώ ε, στη Κλειφόζάτη γιατί δεν απαντήσατε στο συνάδελφο οπότε θα θέσω και πάλι το ερώτημα. Ένα ερώτημα κλειστού τύπου αν θέλετε, στο οποίο μπορείτε να απαντήσετε με ναι ή όχι. Δηλαδή, θα σεβαστείτε το σχετικό ψήφισμα ε, του ε, Κοινοβουλίου, ένα ε, ψήφισμα το οποίο ψηφίστηκε από μια ευρεία πλειοψηφία του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της χρήσης του γλυφοζάτ το ε, η γλυφοζάτη αποτελεί ε, ένα, μια αντιβιωτική ουσία η οποία δεν είναι πατενταρισμένη και η οποία έχει αρνητικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την, την χρήση άλλων εναλλακτικών αντιβιωτικών παρότι έχει ε, θετικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση μικροβίων. Θα ήθελα να μας πει η Επιτροπή πότε θα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα πραγματικά. Κύριος Μπέχα έχει τώρα το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και στο πλαίσιο του τελευταίου διαρθωμένου διαλόγου είχα θέσει ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού. Είχατε, ήσασταν αισιόδοξο, παραμένετε αισιόδοξο και τώρα, αλλά εάν ε, δω τις στατιστικές, τι διαπιστώνω, ότι 5 έως 6 κράτη-μέλη έχουν πραγματικά εφαρμόσει την εθνική του νομοθεσία, την οδηγία. Όμως στις 20 Μαΐου εκπνέει η προθεσμία για την εφαρμογή στην εθνική νομοθεσία. Οπότε ε, προβληματίζομαι και γνωρίζω και στη δική μου χώρα πώς πάνε τα πράγματα στο επίπεδο της εφαρμογής. Ενδεχομένως λοιπόν να προκύψουν προβλήματα στην ε, εφαρμογή της οδηγίας ε, αυτή καθεαυτή. Και υποψιάζομαι ότι τα πράγματα είναι αντίστοιχα και σε άλλα κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν θα ήθελα να μου διευκρινίσετε το εξή. Εάν τα κράτη-μέλη δεν καταφέρουν να εφαρμόσουν την εθνική νομοθεσία, την οδηγία έω την προθεσμία, ποιε θα είναι επιπτώσει, ποια θα είναι τα μέτρα που θα λάβει η Επιτροπή. Θα εφαρμοστεί άμεσα η οδηγία, ναι ή όχι. Ή, εν πάση περιπτώσει, αναλογίζεται η Επιτροπή τα μέτρα τα οποία θα λάβει σε μια τέτοια περίπτωση και από εκεί και μετά και ο κλάδο τι θα κάνει από την πλευρά του των προϊόντων ε, καπνού. Ακούσαμε ότι υπήρξε και μια έκκληση για την ε, παράταση τη σχετική προθεσμία έω τον επόμενο ε, χρόνο. Θα μπορούσατε να μας δώσετε μια πληροφορία σχέση με αυτό. Ο κύριο Φαρία. Ναι. υπήρξε η υιοθέτηση ενό ψηφίσματο σε ό,τι αφορά του ε, περιορισμού τη χρήση τη γλυφοσάτη για τα επόμενα 7 χρόνια και βέβαια πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τα ζητήματα της δημόσιας υγείας. Οπότε, ε, όπως ε, ήδη αναφέρθηκε, υπήρξε υιοθετήθηκε ε, το ψήφισμα σε ό,τι αφορά τη ε, γλυφοσάτη στο πλαίσιο μιας ε, διαφοράς απόψεων σε σχέση με τα, με τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής τη ουσία με βάση μια αξιολόγηση από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη διαφοροποίηση εδώ των απόψεων, οπότε το να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά ε, το, την διάθεση στην αγορά ή όχι του συγκεκριμένου προϊόντος, παρότι αυτό αποτελεί δική μου προσωπική άποψη. Σε ό,τι αφορά την αφορά την τοξικότητα της ε, γλυφοζάτης. Εάν ε, πραγματικά αποφασιστεί ότι αυτό το φυτοφάρμακο είναι τοξικό, εάν διαπιστωθεί αυτό, τι σκοπεύει να κάνει η Επιτροπή σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Και πώς είναι δυνατό η Επιτροπή να έχει προβλέψει ε, ένα χρονοδιάγραμμα τόσο ευρύ ως το 2031. Ε, ενώ έχουν ληφθεί από άλλους φορείς αποφάσεις για τον περιορισμό. Ε, ε, Για το ΣΥΚΑ είναι μία από τις προτεραιότητες ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο, στη Βραζιλία βλέπουμε δημοσιεύματα βάσει των οποίων υπάρχει επιτυχία στην καταπολέμηση της επιδημίας. Έχετε γνώση αυτών των πληροφοριών και τι σκοπεύετε να κάνετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σομέχε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, ε, είχα προβλέψει και εγώ να σας υποβάλω ερωτήματα για την γλυφοσάτη. Στην ε, απάντησή σας είπατε ότι προτίθεστε να ε, χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν για να καταλήξετε συμβαστική λύση και σε αυτό που εσείς εκλαμβάνετε μια λογική απόφαση. Η μοναδική λογική απόφαση είναι να σεβαστείτε την άποψη του Κοινοβουλίου. Διότι ουσιαστικά πρόκειται για το σεβασμό της δημοκρατίας και έτσι θα νομοποιηθείτε στα μάτια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μοναδική απόφαση που συνάδει με την αρχή της πρόληψης είναι να μην δοθεί άδεια για την γλυφοσάτη μέχρι που να έχετε ε, στη διάθεσή σας ανεξάρτητες ε, ε, μελέτες, επιστημονικές μελέτες. Για την TTIP ε, λαμβάνεται αυτή η διάσταση υπόψη ε, στο μέτρο που ξέρουμε πως ε, γεωργικά προϊόντα στην Αμερική έχουν ανησυχητική, ε, ανησυχητικά υψηλή περιεκτικότητα σε γλυφοσάτη. Επίσης, ε, ως προς την πρόσβαση στην ε, τρι θεραπεία για το AIDS. σε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Πολωνία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, είναι ιδιαίτερα περίπλοκη η πρόσβαση λόγω της τιμής. Ε, αφήστε που υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας ε, και στα φαρμακεία και στα νοσοκομεία ε, και στα, νοσοκομ... στα φαρμακεία των νοσοκομείων ε, και στα ιδιωτικά φαρμακεία. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι για την εξασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών. Ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Στάις τώρα. Ευχαριστώ. Είπατε πως ε, ε καλωσορίζεται το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την γλυφοσάτη και Λέτε ότι σα ικανοποιεί το περιεχόμενο. Χαιρόμαστε που μας το λέτε, αλλά τι θα συμβεί. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις υπηρεσίες Επιτροπή ε, και τα κράτη-μέλη. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί ξεκάθαρα για τα κριτήρια μας. Ε, μία επαγγελματική χρήση της ε, γλυφωσάτης, όχι κοντά σε πάρκα, σε χώρους αναψυχή. Αν ζητήσαμε να μα πείτε αν υπάρχουν άλλε μέθοδοι καταπολέμηση των ζυζανίων Επίσης, ε, όχι ε, καμία χρήση, απαγόρευση χρήσης ε, γλυφοσάτης πριν από τη συγκομιδή και ούτω καθεξής. Έχουμε όμως δει δημοσιεύματα στον τύπο για αυτές τις φήμες ότι θα δοθεί προσωρινή αδειοδότηση για 10 χρόνια. Καλωσορίζετε λοιπόν το, το ψήφισμα και δηλώνετε ικανοποιημένο με το περιεχόμενο. Μπορείτε να μα διασφαλίσετε ότι τι επόμενε τρει σε τέσσερι εβδομάδε εσεί προσωπικά θα αναλάβετε δράση, ούτω ώστε να ε, υπάρξει ε, συμμόρφωση με αυτά τα τέσσερα κριτήρια που έθεσε στο ψήφισμά του το Κοινοβούλιο ε, για την πρόταση που θα καταθέσετε στι 18 και 19 Μαου. Διότι πρόκειται για την απόφαση που θα λάβουν τα κράτη-μέλη επί τη βάση τη δική σας πρότασης. Ε, τι σκοπεύετε να κάνετε. Ευχαριστούμε η κυρία Εύη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Θα ήθελα να ε, μιλήσω για την κατάσταση στο νότιο Τιρόλ. Εδώ, εδώ, εδώ πίσω είμαι. Ε, σε αυτή την υπέροχη κοιλάδα στο Μάλις 92% του ε, του, του τοπίου διατηρείται με φυσικό τρόπο, παρόλα αυτά χρησιμοποιούνται ζυζανιοκτώνα. Περισσότερο από ό,τι σε άλλα μέρη της Ιταλίας. Ε, και τι μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει, χρησιμοποιούνται, χρησιμοποιούνται αδιάκριτα αυτές οι ουσίες. δηλαδή σε ποδηλατοδρόμους, σε σημεία όπου κυκλοφορούν τουρίστες, πολίτες, ε, αυτοί που χρησιμοποιούν τα ζυζανιοκτώνα έχουν τον προστατευτικό ρουχισμό και εξοπλισμό, όμως ε, σε πάρα πολύ εκτεταμένες περιοχές ε, χρησιμοποιείται το ζυζανιοκτόνο και εκεί δεν υπάρχει καμία προστασία. 75% των ερωτηθέντων μετά από μια δημοσκόπηση είπαν ότι θέλουν να καταργηθεί η χρήση αυτού του ζυζανιοκτόνου στη συγκεκριμένη κοιλάδα μάλιστα. Θα εισακουστεί λοιπόν ε, η επιθυμία των πολιτών θέλουν να χρησιμοποιηθούν άλλες μέθοδοι ε, καταπολέμησης των ε, ζυζανίων. Θέλουν να χρησιμοποιηθούν παραδοσιακές μέθοδοι. Πώς ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις ανάγκες των πολιτών που ζουν στις παρακείμενες περιοχές, εκεί που χρησιμοποιούνται τα ζενεκτόνα αυτά. Ευχαριστούμε κυρία Γκουντή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Ε, για τα μεταλλαγμένα και τις επιστημονικές εκθέσεις, επειδή περιμένουμε την έκθεση το 2016, το crispr cas ε, που θεωρείται η εφεύρεση του αιώνα θα ληφθεί υπόψη, διότι πρόκειται για εγχειρήσεις ε, που επηρεάζουν το γονιδίωμα και αυτό πέρα από την γεωργία δημιουργεί θέματα ηθικής και υγειονομικά ζητήματα. Επειδή υπάρχουν προθέσεις περιοριστεί η χρήση κυρίω ω προ τα ανθρώπινα έμβρια, θα πρέπει να μα ενημερώσετε για τι προθέσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ρυθμίζετε τη χρήση αυτή τη νέα τεχνολογία για τι διάφορε εφαρμογέ ε, ή θα επιβάλλετε μορατόριο για το γονιδίωμα μέχρι ότου τα υγειονομικά και τα ηθικολογικά ζητήματα να ε, συζητηθούν και να ε, ρυθμιστούν σε επίπεδο κρατών μελών. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γκαρντίνη αλλά ε, υποφέρει από η κυρία Γκαρδίνη και θα τα πω εγώ για εκείνη. Όταν μιλάμε για την υγεία, πολλέ φορέ και όσον αφορά την Ευρώπη και τι ε, ανισότητε. Γιατί λένε ότι έχουμε 86% των ευρωπαϊκών νοσοκομείων που έχουν κάποιε έλλειψει όσον αφορά τα, τα, φάρμακα. Για κάποια πάρα πολύ σημαντικό, όπω α πούμε τα φάρμακα για τι σημαντικέ χημειοθεραπείε. Άρα, τι θα κάνετε, ούτω ώστε να άρετε αυτό το μεγάλο δραματικό πρόβλημα, ε, να, να έχετε κάποιο είδου ε, ευρωπαϊκή αξιολόγηση της τεχνολογίας. Αυτό μας το είπατε. Αλλά θα πρέπει να μην έχουμε τις ε, σχετικές ε, επικαλύψεις, να μην έχουμε τη διασπάθηση των πόρων που γίνεται γιατί έχουμε την Ευρωπαϊκή τα Φάρμακα που πρόσφατα τα παρουσίασε πάρα πολύ στρογγυλά για ε, ένα πιλωτικό πρόγραμμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο, δε διευθυντή τη υπηρεσία είπε ότι έτσι πρόκειται να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε πάρα πολύ σημαντικά φάρμακα για όλη την Ευρώπη. Οπότε, ε, με δεδομένο αυτό, τι θεωρείτε, δεν θεωρείτε κύριε Πίτρο ότι ήρθε η ώρα ούτως ώστε να έχουμε αυτή την ευρωπαϊκή αξιολόγηση των, ε, των ιατρικών τεχνικών, θα κατεβάσετε κάποιο νομοθέτημα προς αυτή την κατεύθυνση και τώρα λέει ο Πρόεδρος, κύριε Σάρπο. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, τον προηγούμενο μήνα παρουσιάσατε την ε, πρότασή σας για τα τρανς ε, λιπαρά. Όμως, δεν έχουμε νομοθετική πρόταση γιατί πρόκειται για μια διαδικασία που θα κρατηθήσει πολύ. Άρα για να μας νομοθετική πρόταση. Πότε θα υποβληθεί από πλευρά σα, Ο κύριος Τόρμαν. Ευχαριστώ. Επίτροπε, μας ε, ενημερώσατε όσον αφορά την ε, οδηγία για το κάλεσμα και είπατε ότι είναι προτεραιότητα η εφαρμογή της οδηγίας και ότι κάνετε ό,τι μπορείτε, ούτως ώστε τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τη σχετική προθεσμία. Μα φτάσαμε σε ένα μήνα, εκπνέει η προθεσμία και δεν βλέπω εύκολα να πετύχει το στόχο. Γιατί στις 8 Απριλίου παραδέχθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μόνο 5 στους 28 πρόκειται να έχουν κάνει ό,τι χρειάζεται και ό,τι προβλέπεται για την επόμενη διετία. Υπάρχει βέβαια και η καπνοβιομηχανία, όμως ξέρετε ότι για την Δανία η εξαγωγή καπνού είναι κάτι πολύ σημαντικό για την οικονομία μας. Και έχουμε μια εταιρεία που έχει 140 εργαζομένους. Τι με το άρθρο 11. Δύο είναι τα πιθανά σενάρια. Διπλή προετοιμασία των συσκευών, ε, διπλή προσπάθεια και άρα έχουμε αύξηση των εξόδων επιμελητίας. Έχουμε δύο θεσμικά όργανα για να εφαρμόσουν την κοινοτική νομοθεσία. Θα κάνετε αυτά τα οποία πρέπει. Νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπόρεσε μέχρι τώρα να κάνει ό,τι έπρεπε. Δεν ξέρω. Ανησυχώ για το τι θα κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ο κύριος Εκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Επιτροπέ Αντριουκάητης. Σας ευχαριστούμε καταρχήν για τη δυνατότητα που μας δίνετε να κάνουμε αυτό το διάλογο σήμερα μαζί σας. Επιτρέψτε μου να εκφράσω όμω τις αμφιβολίες μου σε ό,τι αφορά δύο πρόσφατες πρωτοβουλίε ε, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, καταρχήν, σε ό,τι αφορά την πρόταση για τον ψευδόργυρο και δεύτερον σε ό,τι αφορά την Παρασκευή ε, φυτοφαρμάκων, ε, λιπασμάτων, συγγνώμη. Ε, ο ψευδάρκιος και διάφορες ε, φωσφορικές ενότητες μπορούν ε, να χρησιμοποιηθούν όπως και το κάδμιο και το νικέλιο για την παρασκευή τέτοιων προϊόντων και ακριβώς για αυτόν τον λόγο ο κανονισμός θέτει συγκεκριμένους περιορισμούς σε ό,τι αφορά την χρήση βαρέων μετάλλων στα λιπάσματα ώστε να αποφευχθεί ακριβώς και το πέρασμά τους μέσα στην τροφική αλυσίδα. Ε, και μάλιστα τα όρια για το κάδμιο ε, προβλέπονται να μειωθούν σε τρία χρόνια. Ε, Σα ρωτάω λοιπόν, ε, σε σχέση με τον Ψετάκηρο, πότε προβλέπετε να γίνει κάτι τέτοιο. Όπω λέμε, γίνονται συστηματικέ προσπάθειε μείωση τη χρήση γενικότερα του ψευδαργύρου, αλλά από την άλλη πλευρά ε, επιτρέπουμε τη χρήση ε, ε, φωσφορικών ενώσεων στα λιπάσματα, τα οποία βέβαια μπορούν να περιέχουν πολύ μεγάλες ποσότητες ψευδαρκύρου. Οπότε, γιατί οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ είναι κατά κάποιο τρόπο αντιφατικές μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Πέτρελε. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της γλυφοσάτης, να πούμε ότι κάποιοι έχουν ε, αναφέρει ότι δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικέ. Ε, γενικότερα δεν υπήρχαν εναλλακτικέ όταν ζούσαμε κάποτε σε μη δημοκρατικά καθεστώτα. Έκτοτε υπάρχουν εναλλακτικέ. Θα ήθελα να μας πει η Επιτροπή τι θα κάνει σχέση με αυτό το ζήτημα, ούτως ώστε να μην παραμείνουμε όμοιροι της χημικής βιομηχανίας. Και εδώ βέβαια δεν Αναφέρομαι μόνο για του αγρότε όσο ομίλου τη χημική βιομηχανία. Από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, τα τρανς λιπαρά θα παραμείνουν στα πιάτα μας αν θέλετε για, ένα, ε, ε, για, αρκετό ε, για αρκετό χρονικό διάστημα από εδώ και στο εξή. Οπότε πότε θα υπάρξει μια συγκεκριμένη πρόταση από την Επιτροπή. Επίση, ε, σε ό,τι αφορά ε, ε, ε τι προτάσει τη Επιτροπή, σε ό,τι αφορά του πυλώνε κοινωνική προστασία, αναφέρεται εκεί ότι και η προστασία τη υγεία θα περιλαμβάνεται. Οπότε, ποιο θα είναι ο ρόλο που εσεί θα αναλάβετε σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή η κοινωνική πτυχή θα αποτελέσει τμήμα και των πολιτικών ε, προστασίας της υγείας μέσα και στο, ε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ε, έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε μια ε, συνεδρία σε ό,τι αφορά τον καρκίνο του δέρματος και αναφέρθηκε ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξει δραστηριοποίηση, δραστηριοποίηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε, τι έχετε κάνει για αυτή την προετοιμασία, ειδικότερα και σε ό,τι αφορά και την οδηγία 37. Από εκεί και μετά, ένα ακόμα ε, ερώτημα σε ό,τι αφορά τη μικροβιακή αντοχή. Και εδώ διαρωτόμαστε ποιε είναι εναλλακτικέ ε, που έχουμε στη διάθεσή μα. Θα θέλαμε να υπάρξουν εναλλακτικέ μέθοδοι δηλαδή σε ό,τι αφορά το, τι μπορούμε να κάνουμε τόσο ώστε να βελτιώσουμε και την ε, υγεία των ανθρώπων και των ζώων φυσικά. Ε, θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, Κάντεμπαχ. Ε, ευχαριστούμε. Ε, θερμά εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Πέτρελε γιατί χωρίς να έχουμε συζητήσει μεταξύ μας ε, προηγουμένως ε, με κάλυψε σε μεγάλο βαθμό στα ερωτήματα μου. Δηλαδή κατά τα τελευταία έτη αναφέρθηκε ε, επανειλημμένα το ζήτημα της πρόληψης, της επένδυσης στη δημόσια υγεία και ειδικότερα το ζήτημα της αλληλεγγύη 68 ότι θα πρέπει, δηλαδή, συγγνώμη, το άρθρο 68 ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται το ζήτημα της υγείας στο πλαίσιο όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διάσταση της υγείας, αλλά βλέπουμε ότι δεν βλέπουμε τίποτα ε, πια σήμερα σε σχέση με αυτές τις πολιτικές υγείας, δεν βλέπουμε κάτι να αναφέρεται προς την κατεύθυνση της πρόληψης, οπότε πραγματικά είναι σημαντικό να επιμείνουμε σε αυτή την αξίωση. Δηλαδή το ζήτημα ε, της υγείας συμπεριλαμβάνει και επενδύσεις στον χώρο της υγείας. Για παράδειγμα ε, health literacy και άλλα αντίστοιχα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να περιληφθούν στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγηθούμε στην κατάσταση που είχαμε και στο παρελθόν. Δηλαδή μιλάμε συνέχεια για την νομοθεσία, ότι χρειαζόμαστε περισσότερη νομοθεσία, αλλά τελικά βλέπουμε ότι η εφαρμογή της στην πράξη δεν είναι καλή, δεν είναι συνεπής, όπως συμβαίνει για παράδειγμα και με την οδηγία για τα προϊόντα ε, καπνού. Και από εκεί και μετά έχουμε υπερβολικά χρονοβόρες ε, αξιολογήσεις αντικτύπου, οπότε πραγματικά και σε σχέση με το σχέδιο δράσης σε ό,τι αφορά την ε, ε, πρόληψη για τις μακρόχρονες ασθένειες υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και θα πρέπει να δούμε να υπάρξουν τα κατάλληλα ε, εργαλεία και να δοθεί κατάλληλη προτεραιότητα, γιατί μέχρι στιγμή βλέπουμε ότι σε αυτέ τι ε, πολιτικέ και ε, από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την πλευρά των κρατών μελών δεν αποτελεί ζήτημα προτεραιότητα η υγεία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που ακόμη δεν σχολιάστηκε. Το ευζήν των ζώων. Μπροστά σας είμαι. Η βιομηχανία χειροκρεατός ε, γίνονται συζητήσεις στην Επιτροπή Γεωργίας για την κρίση ε, σε αυτή τη βιομηχανία ε, και στη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων επίσης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι βιώσιμη επιχείρηση των εκτροφέων και των γεωργών με την νέα νομοθεσία. Είναι πάρα πολύ κακή η κατάσταση για το χείριο κρέας και τα γαλακτοκομικά. Πρέπει να, εμείς να φροντίσουμε ώστε να είναι βιώσιμη η επιχείρησή τους. Με την TTIP ε, πώς ακριβώς σκοπεύετε να το κάνετε αυτό. Τι θα κάνουν τόσες οικογένειες, ε, διότι ε, πολεμάνε κατά των πολυεθνικών που έχουν χιλιάδες ζώα ε, με πολύ μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο. Ευχαριστούμε. Η κυρία Καβεσόν. Πρόεδρε, μας είπατε ότι έγινε άτυπο Συμβούλιο Υγείας του Άμστερνταμ. Νομίζω ότι τα συμπεράσματα είναι πάρα πολύ καλή αφετηρία έλεγαν για το πόσο σημαντική είναι η φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη. Λέγανε για το ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία σε αυτόν τον κλάδο. Ε, θεωρούσαν ότι δεν είναι βιώσιμη κατάσταση για τα κρατημέλη και ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Ε, ε, βέβαια είπαν τελικά ότι πιο σημαντική είναι η βιομηχανία από τον κόσμο και αυτό το είπαν ακριβώς έτσι λέγοντας ότι θα πρέπει να δουν την τιμολογική πολιτική, να δουν τις δαπάνες, ε, κόστος και προσθέμενη αξία. Επίσης ε, λέγαμε για τις καταχρήσεις στο σύστημα των ε, έβρεση τεχνιών και ακριβώς όπως σας είπα είναι αφετηρία αυτό το έγγραφο. Λέει και άλλα πράγματα. Αλλά σημαίνει ότι είναι αποφασισμένα τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν και επίσης ζητείται μία λύση α, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης να υπάρξει και ανταλλαγή πληροφοριών. Όλα αυτά αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο, οπότε εμείς δεν είναι δυνατόν να ε, παρακάμψουμε αυτά τα οποία συζητήθηκαν ή επίσης ο καθορισμός των τιμών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας και επίσης θέλω να μου επαναλάβετε ότι στρατεύεστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο επόμενος είναι ο κύριος Πολούτσι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε με ευρεία πλειοψηφία ζητήσαμε ε, την εφαρμογή του άρθρου 4 του κανονισμού του 2006 και το είπαμε στην νομική επιτροπή και στην Ολομέλεια επανειλημμένα ότι θα πρέπει να προσεχθεί η ε, υγεία μέσω σωστών υγιεινών ειδών διατροφής και θα πρέπει να υπάρχουν είδη διατροφής υψηλής ποιότητας. Και επίσης θα πρέπει να υπάρχει ε, ενημέρωση του καταναλωτή με σωστή διαφήμιση και να σταματήσει να, υπάρχει αυτό το χάος το, των ε, ειδών διατροφής χαμηλής ποιότητας. Τι θα κάνετε γι' αυτό. επόμενος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Επίτροπε που δίνετε απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματά μας. Ε, επανέρχομαι στο ζήτημα της γλυφοζάτης. Μας είπατε ο ίδιος ότι σε ε, συντονισμό με τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιτύχουμε κάποια πρόοδο, να φτάσουμε σε μια λύση ε, και γίνεται λόγος για άδειε χρήσης διάρκειας 10 ετών. Θα ήθελα να μου επιβεβαίωσε ότι αν μιλάμε πραγματικά για 10 χρόνια ή όχι. Και επίσης υπήρξε μια πρόταση ε, επανειλημμένα από την πλευρά κάποιων κρατών μελών, ειδικότερα από την πλευρά της Γερμανίας, σε ό,τι αφορά το ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τη χρήση ε, της ε, γλυφοζάτης και ειδικότερα σε συγκεκριμένες περιόδους πριν ακριβώς από τη συγκομιδή, ε, μετά από την, και την απαγόρευση της χρήσης από μη επαγγελματίες και αυτό γιατί αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα ότι δηλαδή η γλυφοζάτη χρησιμοποιείται από μη επαγγελματίε ε, στη Γερμανία. Ε, και μετά η χρήση τα μεβαμένων, για παράδειγμα, δηλαδή συμπληρωματικών ουσιών, ε, οι οποίες ενδεχομένω θα πρέπει να απαγορευτούν μαζί με τη γλυφοζάτη. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε εάν πράγματι περιλαμβάνονται όλα αυτά στις δικέ σας σκέψει. Ευχαριστώ, λέω πρόεδρο, κυρία Πούτλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Ξέρετε ότι ε, πολύ υψηλό κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι βακτηριοδικέ μολύσει. 250.000 εκρούσματα φέτο και για το 2014, σε σχέση με το 2014 είναι πολύ πιο ανησυχητική η κατάσταση. Θέλω να ξέρω αν προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιήσει την νομοθεσία για τα καμπυλοβακτηρίδια σε σχέση με την επεξεργασία του, ε, των πουλερικών και τις απολυμάνσεις. Ευχαριστούμε ο κύριος Τσόφολη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, εγώ θέλω να επενέλθω στο ζήτημα ε, ε, της ετικετοθεσίας για την προέλευση όσον αφορά τα επεξεργασμένα κρέατα και κυρίως το, το βόλιο. είδαμε την πρωτοβουλία της Γαλλίας και είδαμε τα δύο ψηφίσματα τα οποία είναι, υπέρ του, είναι υποχρεωτική η ετικετοθεσία. Τα ψηφίσματα τα δικά μας του Κοινοβουλίου. Οπότε εγώ θέλω να σταθώ στο ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει και έτσι να υπάρξει εγγύηση διαφάνειας για όλη την διαδρομή στην νέα αγορά. Μην έχουμε ε, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπο, λέει κυρία Σκαλντεμός. Μας είπατε ότι θα νομοθετήσετε ούτω ώστε να υπάρχουν λιγότερα τρανς λιπαρά στα είδη διατροφής. Όμως, το σημαντικό για το οποίο μίλησαν πολλοί συναδελφοί είναι η γλυφοσάτη. Από ό,τι γνωρίζουμε, πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό προβληματισμό όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου. Η υπηρεσία ΕΦΣΑ έχει κάποιες προτάσεις για οριακές τιμές. Εσείς μπορείτε να διευρύνετε την ε, εντολή προς την ΕΦΣΑ ούτως ώστε να δείτε τα πράγματα ε, πιο σφαιρικά. Αξίζει περισσότερων πόρων. Μπορείτε να την πληκοδοτήσετε Ευχαριστούμε, λέει ο κύριος Λαβία. Και τώρα σκητάλη στον κύριο Επίτροπο για τις απαντήσεις. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αλλά ίσως μπορείτε κι εσείς να συμπυκνώσετε τις απαντήσεις Thank you very much All questions... Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα τα ερωτήματα. Και καλό θα ήταν να ζητήσω από την ομάδα μου να συνοψίσει τα ερωτήματα και μετά να λάβετε και διεξοδικότερες απαντήσεις, διότι δεν γίνεται να απαντήσω τώρα ε, ξεχωριστά σε όλα τα ερωτήματα. Μπορώ να κάνω μία σύνοψη για τη γλυφοσάτη και όλα τα συναφή ζητήματα. Ξαναλέω. συζητάμε αυτά τα θέματα με τα κράτη-μέλη. Συμμετέχω σε αυτές τις συζητήσεις και λαμβάνω υπόψη το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του οποίου το περιεχόμενο εγκρίνω, ξαναλέω, πρέπει όμως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συζητήσουν ε, σε επίπεδο ε, διπηρεσιακό στην Επιτροπή, με τα κράτη-μέλη, με το Κοινοβούλιο, σε επίπεδο σώματος επιτρόπων ε, με τους εμπλεκόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Όλοι θα πρέπει να συζητήσουμε για αυτά τα ζητήματα. Φυσικά ποιος θα ήταν κατά της αυστηρότερης ρύθμισης Και ποιος θα ήταν κατά του να λαμβάνουμε υπόψη όλα αυτά, όλα αυτές τις διαστάσεις του ζητήματος για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Φυσικά και για τη βιομηχανία είναι πολύ ε, ωφέλιμο να υπάρχει μια αυστηρότερη νομοθεσία. Ο ΕΦΣΑ ε, έχει ε, επιλεχθεί του ε, ζητήματος, ε, ε, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το ΙΑΡΚ, είναι διαφορετικός μηχανισμός, χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους. Ε, παραδείγματος χάρη, το κόκκινο κρέας είναι καρκινογενές. ορίστε, έκθεση από την ΙΑΡΚ. Γιατί δεν αγχωνόμαστε γι' αυτό. Και το ίδιο είπε και για την γλυφοσάτη γιατί μιλάει για κίνδυνο η ΑΡΚ. Όμως ε, για την αποτίμηση κινδύνου έχουμε αρμόδιο οργανισμό, τον ΕΦΣΑ. Ναι, φυσικά χρειάζεται περισσότερους πόρους ε, για να κάνουν αξιολόγηση, αλλά δική μας και δική σας δουλειά είναι. Όλοι εμείς ε, αποφασίζουμε μετά από ευρεία διαβούλευση για τον προϋπολογισμό και τους πόρους που θα θέσουμε στη διάθεση του ΕΦΣΑ. Ωραία, συμφωνώ μαζί σας. Καλό θα ήταν να έχουμε το 100% των αναγκών μας σε δημοσιονομικές προβλέψεις ε, ε, και να μην βασιζόμαστε ε, στην βιομηχανία όμως. Δεν μπορώ εγώ μόνος μου να πάρω αυτή την απόφαση. Φυσικά χρειαζόμαστε ένα μερόληπτο οργανισμό αξιολόγησης, όμως πρέπει να καταλάβετε πως ε, πρέπει να κατοχυρώσουμε και την απόλυτη διαφάνεια μέσα στο πλαίσιο της ένομης τάξης και του, ε, των ρυθμιστικών διατάξεων που μεταξύ άλλων ενέκρινε και το Κοινοβούλιο. Εάν δεν υποστηριχθεί η ανανέωση της άδειας, Ξέρετε, τα κράτη-μέλη μπορούν να καταργήσουν την ε, άδεια θέση εμπορία της γλυφωσάτης. Μιλήσαμε για την Τσεχία, τη Γερμανία, την Πολωνία. Μην ξεχνάμε ότι μπορούν και τα ίδια τα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν την κατάσταση και ε, ε, να καταργήσουν τη χρήση της εγκλυφωσάτης στην περίοδο πριν τη συγκομιδή. Φυσικά χρειάζεται ενημερωτική εκστρατεία χρειάζονται δράσεις ε, ε, ενημέρωσης ε, των χρηστών σε επίπεδο κράτους μέλους, μη μικρών κοινωνίας των πολιτών. Και για να γίνουν αυτά θα πρέπει να επικρατήσει η απόλυτη διαφάνεια, ούτως ώστε να βελτιώσουμε την ασφάλεια των τροφίμων και τα πρότυπα δημόσιας υγείας. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει καμία αντίφαση τα λεβαμίνες. Ε, είπατε ναι, να καταργηθεί. Φυσικά μπορούμε και θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί και άμεσα θα έπρεπε να κάνουμε μία βιοπαρακολούθηση και αξιολόγηση των στοιχείων. Αλλιώς θα απολέσουμε την αξιοπιστία μας. Και φυσικά θέλω να γίνουν αυτές οι συζητήσεις πρωτού αναλυφθεί κοινή δράση. Ό,τι μπορώ να κάνω θα το κάνω και τα κράτη-μέλη θα πρέπει αντίστοιχα να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους. Για την χρήση αυτών των προϊόντων ε, μην ξεχνάμε ότι είναι εθνική αρμοδιότητα όταν μιλάμε για συγκεκριμένα προϊόντα. Οπότε την ίδια κατεύθυνση ακολουθούμε. Στο ίδιο στρατόπεδο είμαστε. Μην θέλουμε ότι κάποιοι είναι φίλοι και άλλοι εχθροί της βιομηχανίας. Καμία σχέση. Δεν ευσταθεί αυτό. Στο ίδιο στρατόπεδο με σας είμαι. Για τα καμπυλοβακτηρίδια είναι, είναι δύσκολο το πρόβλημα αυτό. Βλέπουμε τα στοιχεία και προκύπτει ότι πρέπει να για τα πρότυπά μας ε, σε όλη την αλυσίδα να, ενδεχομένως να κάνουμε διαρκή αξιολόγηση διότι είναι πάνω από 200.000 τα κρούσματα κάθε χρόνο. Και οι κτηνίατροι διαρκώς συζητάνε μαζί μας για την αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου και θέλουμε αυστηρότερη νομοθεσία, νέα μέσα για τον έλεγχο. και ε, είναι σοβαρές συζητήσει ε, που γίνονται διότι δεν έχουμε στα χέρια μας ε, τα ελεγκτικά μέσα για να παρακολουθούμε τη διαδικασία για να καταπολεμήσουμε την επιμόλυνση με κάμπυλοβακτηρίδια. και ε, να δούμε κατά πόσο ε, έχουν μολυνθεί τα κρέατα. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα το οποίο πρέπει επίσης να ζητήσουμε με τους ειδικού για τον καπνό. Ε, για τα εφαρμοστικά μέτρα. Εάν κάποιο κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με τις νομικές του υποχρεώσεις, αμέσως θα εκκινήσουμε τη διαδικασία επιπαραβάση. Δεν είναι χώρα καμία αμφιβολία. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο το μήνυμά μας. Κανέ, καμία, κανένα συμβασμός, ε, καμία υποχώρηση για τον καπνό. Ξέρω ότι δυσκολεύονται κάποιοι διότι θέλουν οι τελικά απόφαση να λαμβάνονται στο κοινοβούλιο. Στη Τσεχία, στη Ρουμανία, συζητάω ε, με βουλευτές ε, στην Πορτογαλία Θέλω να είμαστε αποτελεσματικοί και να, ε, για τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία να ψηφιστούν ε, τα απαραίτητα μέτρα. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Ξέρω προσωπικά, από προσωπική εμπειρία, πόσο καταστροφικό είναι το κάπνισμα. τα κτηνιατρικά μέτρα, ναι. Πιέζω τα κράτη-μέλη να δράσουν σε σχέση με τα κτηνιατρικά φάρμακα και να προχωρήσουμε συζητήσει σε επίπεδο συμβουλίου. Θέλω και πάλι να τονίσω ότι θα πρέπει να επισπεύσουμε το ταχύτερο δυνατό να ληφθεί μια απόφαση και και να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να συνταχθούν τα κράτη-μέλη με το Κοινοβούλιο για να προχωρήσουμε. Για τα καινοτόμα φάρμακα και τη βελτίωση της πρόσβασης στις θεραπείες. Βεβαίως. Πολύ σημαντικό ε, ε πολύ σημαντικό τομέας ε, για μένα. Είμαι σε διαρκή επαφή με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Είναι πολύ καλό αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Μόλις τώρα ξεκίνησε και θα δούμε ποια αποτελέσματα θα έχει σε μισό χρόνο από τώρα. Ενθαρρύνουμε πάντως τα κράτη-μέλη για να ε, πιέσουν από πλευρά τους, πλευράς τους για την τεχνολογία στον τομέα της υγείας και την αξιολόγηση. Υπάρχουν ε, σχέδια για το 2017 για να καταθέσουμε μια πρόταση ε, νομοθετικού περιεχομένου, την πρότασή μας πρώτα βέβαια στο Σώμα των Επιτρόμων και μετά στο Συμβούλιο. Πρώτα πρέπει να γίνει η αξιολόγηση ε, του προγράμματος με κίνητρα σε διάφορους τομείς και τα τελικά αποτελέσματα θα ε, ευελπιστούμε να τα παρουσιάσουμε το 2017. Ξεκινάει η μελέτη αντικτύπου τώρα. για την ευμερία των ζώων. η κατάσταση με τους γεωργούς βεβαίως. Χείριο, κρέας, ε, γαλακτοκομικά προϊόντα ε, αντιμετωπίζουν σοβαρότατες δυσκολίες ε, και ε, έχουμε και το πρόβλημα της παγόρευσης από πλευράς Ρωσίας Φυσικά, σταδιακά πρέπει να εφαρμοστούν τα πρότυπα, ακολουθώντας μια γενική κατεύθυνση και δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές, δημιουργώντας ε, φόρα συζητήσεων, διότι είναι πολύ περίπλοκη η κατάσταση τόπου όπως ξέρετε. Δεν ισχύει η ίδια κατάσταση σε όλες τις χώρες. Ε, κάποιες έχουν προχωρήσει περισσότερο από άλλες. Κάποιες χώρες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Χρειάζεται εξισορρόπηση πάντως. Χρειάζεται μια βάση κοινή για την ευημερία των ζώων, για μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή πρακτικών και για να ενθαρρύνουμε τους γεωργούς και εκτροφείς να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση. Από νομικής πλευράς πάντως, μέχρι το τέλος του 2017 θα μπορέσουμε να έχουμε εκπληρώσει τις νομικές υποχρεώσεις μας για να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες αγοράς. Για το ψευδάργυρο. Ε, υδράργυρο. Ε, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας ενημερώσω διότι δεν ε, κατέχω ε, το ζήτημα. Ε, για τα λοιπάσματα είναι τρεις οι συναρμόδιοι επιτροποί, οπότε θα μεταφέρω τα ερωτήματά σας στους συναδέλφους. για την ε, τεχνολογία, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για τις νέες θεραπείες, για τους ιστούς και για τα κύτταρα και για τις θεραπείες που σχετίζονται με το αίμα. Ε, έχουμε όντως την έκθεση και το ζήτημα είναι αν είναι σαφής η προσέγγιση ούτως ώστε να έχουμε καινοτόμες θεραπείες για χρήση κιτάρων και ιστών. Υπάρχουν διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις για την αποζημίωση των δωρητών και ε, συντρέχει ανάγκη για επαρκή προστασία των δωρητών. Είναι πρόωρο το ζήτημα, δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση προτού γίνει επισκόπηση της κατάστασης ε, θα ξεκινήσει η αξιολόγηση του νομικού πλαισίου για τα κύτταρα και τους ιστούς στο προς τα τέλη του 2016. Για την ετικετοθεσία τα είπαμε, μην τα ξαναπώ. Τι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η έκθεση. Για το που γίνεται διευθυνσιακή διαβούλευση ακόμη. Δεν έχουμε και χρόνο. Εγώ πάντως ε, είμαι στη διάθεσή σας. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες... Και διμερός αν θέλετε να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα λεπτομερέστερα. Thank you very much for your And then uh, now we can uh, close. Uh... Ευχαριστούμε που τώρα μπορούμε να ολοκληρώσουμε μετά από αυτή την τόσο μακρά συζήτηση. Οπότε μπορούμε επί να μπορούμε στο επόμενο σημείο τη ημερησία διατάξεω. Έχουμε τον ε, κύριο Ανδρουλάκη. Ευθύνη αποζημίωση και χρηματοοικονομική ασφάλεια για τι υπεράκτητε δραστηριότητε. Ευθύ αμέσω έχει το λόγο ο κύριο ε, εισηγητή. Παρακαλώ συνάδελφε, λέει ο πρόεδρο, ησυχία. Γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε τι εργασίε μα. Έχετε το λόγο. Συνάδελφοι, πριν ε, περίπου 6 χρόνια, στι 20 Απριλίου του 2010, έγινε η έκρηξη στην πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου Deep Horizon στον κόλπο του Μεξικό. Το ατύχημα αυτό, ίσως το μεγαλύτερο και πιο κοστοβόρο, μέχρι σήμερα οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της προτείνει να αναμένουμε την εφαρμογή της οδηγίας πριν προβεί σε καινούργια νομοθετική πρόταση. Διαφωνούμε σε αυτό το σημείο με την Επιτροπή. Όπω αναφέρω και στην νομοδότηση, ήδη σημαντικό αριθμό υπαράκτιων εταιριών και εγκαταστάσεων είναι πιθανό να αυξηθεί στο μέλλον. Η αύξηση αυτή αναμένεται να σημειωθεί κυρίω στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, όπου οι παράκτιε χώρε δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία ούτε την εμπειρία των χωρών τη Βορείου Θαλάσσου στην αντιμετώπιση τέτοιων ατυχημάτων. Για τον λόγο αυτό θεωρώ αναγκαία την ανάπτυξη του κατάλληλου νομικού πλαισίου το συντομότερο δυνατόν. Πρώτα πρέπει να ασχοληθούμε με τον τομέα τη πρόληψη. Πιστεύω ότι οι πιθανέ ποινικέ ευθύνε θα ευαισθητοποιούσαν του υπευθύνου ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό το λόγο ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την προσθήκη τη παρούσα οδηγία στην οδηγία για το περιβαλλοντολογικό έγκλημα. Ακόμη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα ατύχημα πιθανότητα θα επηρεάσει περισσότερο από ένα κράτη-μέλη. Καθώ ο κανονισμό Ρώμη 2 προβλέπει ότι εφαρμόζεται η νομοθεσία του κράτου όπου επήλθε η ζημιά ανεξαρτήτω του πού συνέβη το ατύχημα. Υπάρχει περίπτωση κάποιοι πολίτε που έχουν υποστεί ζημιά να βρεθούν σε χειρότερη θέση από του γείτονέ του σε άλλο κράτο μέλο που υπέστησαν ζημιά από το ίδιο ατύχημα. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να θεσπίσουμε αυστηρού περί ευθύνη κανόνε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε θα έχουν εύκολη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Τομεί που πλήττονται άμεσα από τέτοιου είδου ατυχήματα, όπω είναι η αηλία και ο τουρισμό, ο παράκτη τουρισμό, πρέπει να την χάνουν ιδιαίτερη προστασία και στο πλαίσιο αυτό καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το παράδειγμα τη Νορβηγία. Τέλο, πιστεύω ότι ίσω πρέπει να εξετάσουμε την ανάγκη κάποιων κοινών κανόνων στον τομέα τη οικονομική ασφάλεια, ιδιαίτερα σχετικά με του μηχανισμού και τα μέσα χρηματοοικονομική κάλυψη και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται από τι εθνικέ αρχέ αδειοδότηση το ύψο των πιθανών ζημιών από ατύχημα. Να υπάρχει ευελιξία ώστε τα κράτη-μέλη και οι φορεί εκμετάλλευση να επιλέγουν το καλύτερο ή τα καλύτερα ανάλογα με την περίπτωση. Άλλωστε, η συγκεκριμένη αγορά είναι ακόμη υπό ανάπτυξη. Όμω ο τρόπο με τον οποίο καταλήγουμε στο ασφαλιζόμενο ποσό και η πιστοποίηση ότι υπάρχει απαραίτητη εξασφάλιση πρέπει να βασίζεται σε κοινού ευρωπαϊκού κανόνε. Θέλουμε να ενισχύσουμε τι προσπάθειε εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών κοιτασμάτων που μπορούν να έχουν θετικά αποτελέσματα και στο ζήτημα τη ενεργειακή ασφάλεια. Όμω αυτό δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση ει βάρο του περιβάλλοντο, χωρί να υπολογίζουμε πιθανέ συνέπειε σε ευαίσθητου οικονομικά τομεί όπω είναι η αλληλεία και ο παράκτητο τουρισμό. Αναμένω τα σχόλιά σα και τι παρατηρήσει σα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Uh, and... Uh, Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πατησέλα από το ΕΛΚΑ μου είπε να πω τα δικά του. Το θέμα της ευθύνη, όσον αφορά την ε, αποζημίωση ε, για τις πράκτες εργασίας του πετρελαιοκυρικού αερίου τις τελευταίες χρονιές είναι θέμα ευρεία συζήτησης σε εθνικό, τοπικό και διεθνές επίπεδο. Το 85% του και το 65% του φυσικού αερίου στην Ευρώπη προέρχεται από τέτοιες εργασίες υπεράκτιες. Και ε, αυτό γίνεται στην Μαύρη Θάλασσα και αλλού. Είναι κάτι επομένως πάρα πολύ σημαντικό την ενεργική πολιτική. Έχουμε ήδη 1.300 εργασίες ε, στην ε, Ευρώπη. Οπότε και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ θετική η προσπάθεια και το έργο του συναδέλφου Άνδρου Λάγκη που θέλει να υπάρξει ρύθμιση και εναρμόνιση των όσων είχε στα κράτη-μέλη. Όσον αφορά την αποζημίωση για ασφάλεια σε αυτές τις εργασίες. Και έτσι νομίζω θα υπάρξει περισσότερη ομοιογένεια. Οπότε θα αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό. Αλλά θα πρέπει να προσέξουμε και το περιβάλλον αλλά και τις ανάγκες των Ευρωπαίων. Να υπάρξουν οι χρηματοοικονομικές εγγύησεις, να καλυφθούν ε, αυτοί οι κίνδυνοι από την ε, διαχείριση των εργασίων αυτών και να δούμε τι θα γίνει με αυτή την αστική αποζημίωση και αστική αθήνη Έχουμε επίσης ε, και ανεπάρκεια προς το παρόν των εγγυήσεων οπότε θα πρέπει να αρθούν αυτά τα κενά στο δίκαιο και νομίζω ότι η πρόσφατη οδηγία για την ε, ασφάλεια της πρακτικής εργασίας ε, δεν έχει τύχει ακόμη πλήρους εφαρμογής. Άρα θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική και επίσης να υπάρχει εγγύηση για προστασία του περιβάλλοντος αλλά επίσης να εξασφαλίσουμε την ε, ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Αυτά από πλευράς του κυρίου Πατριτσέλο. Φαρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ανδρουλάκη για τη δουλειά που έκανε για αυτή την έκθεση. Ε, στο, στην πλατφόρμα Deepwater Horizon το 2010 και το σοβαρότατο ατύχημα που συνέβη εκεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε την κατάρτιση ενός νέου πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος, ε, για τις υπεράκτες επιχειρήσεις για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ε, στις οδηγίες 2013-30 ε και μετά έχουμε την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη και την οδηγία για την αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου που συνδυάζονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτών των επιράκτων επιχειρήσεων ε, θα πρέπει να υπάρχει μια μοναδική διαδικασία αξιολόγησης ε, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αξιολόγηση κινδύνου, κατάρτιση του προσωπικού, ε, ικανοποιητικοί μηχανισμοί οικονομικής αποζημίωσης για τα ατυχήματα ή για τα θύματα υπεράκτειας μόλυνσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επεκτείνει τις ρυθμίσεις που υπάρχουν για την περιβαλλοντική και την αστική ευθύνη και να ταξινομήσει τα αποτελέσματα ενό σοβαρού επιτυχήματο ως προς τις ε, αξιόπινες ε, πράξει. Ε, υπάρχει σοβαρή ανησυχία σε σχέση με τη δράση Ευρωπαϊκή Επιτροπή που χρειάζεται για την, δράση, την αποτρεπτική δράση σε σχέση με την οδηγία για την υπεράκτεια ευθύνη. Πριν ξεκινήσει η δίωξη για τι αξιόπινες πράξεις προκύπτουν από τέτοια ατυχήματα. Η ποινικοποίηση ορισμένων συμπεριφερών έχει αποτρεπτική ισχύ και παρόλα αυτά δεν υπάρχουν όμως αποτελεσματικά ε, μέτρα ε, αποτρεπτικά και μπορούν μόνο να επισύρουν ε, ένα υψηλό κόστος για την προστασία της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Μήπως θα ήταν προτιμότερο να προκρίνεται μεγαλύτερη διαφάνεια και παρακολούθηση της κατάστασης ούτως ώστε να εφαρμόζεται καλύτερα η οδηγία για την υπεράκτη ευθύνη διότι έχουν εντοπιστεί κενά και αμφισημίες μέσα σε αυτή την οδηγία και θα πρέπει να διορθωθούν ε, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ε, που ε, για την αλία, για τον ορισμό ενδεχομένως να είναι σοβαρότατες οι επιπτώσεις αυτών των ατυχημάτων. Οι φορείς εξερεύνησης, παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πρέπει να λαμβάνουν πολύ περισσότερα προληπτικά μέτρα κατά τη γνώμη μου. Και επίσης, όπως είπε και ο εισηγητής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρειάζονται εργαλεία για οικονομική εγγύηση, για τις ζημιές με μεγάλης κλίμακας, ε, ακόμη δεν είναι ικανοποιητικό ο μηχανισμός. Χρειάζεται επίσης σε περιοριστικό πλαίσιο για την αστική και ποινική ευθύνη που υπάρχει σε, προς το παρόν σε κάποια κράτη-μέλη, διότι ενδεχομένως να μην υπάρχει η κάλυψη των ζημιών. Θα υπάρχει ε, τομέας ε, ελέγχου από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μελλοντικές παρεμβάσεις σε περίπτωση που προκύπτει αστική και ποινική ευθύνη. Αυτά, Πρόεδρε, προσβλέπω στην συνεργασία με τον τον εισηγητή και τους κοιόδης. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την γνωμοδότησή του. Πρόκειται να συνεργαστούμε για τις τροπολογίες. Εγώ θέλω να σταθώ στο σημεία. Έχουμε τον 230 του 13 και εκεί μιλά για τα θέματα των ατυχημάτων των σοβαρών, πώς μπορούν να περιοριστούν οι συνέπειες του άρθρου δύο Μιλά για περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών και θανάτων. Αυτό αφορά όχι το περιβάλλον, τα πρόσωπα. Οπότε βεβαίως και είναι αλήθεια ότι μπορεί να υπάρχουν πολύ σοβαρά ατυχήματα και πέραν των προσώπων να έχει παραβλαβεί σοβαρά το περιβάλλον. Οπότε ε, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στο φυσικό περιβάλλον, να υπάρχει βλάβη στην ε, ε, πανίδα και υπάρχουν κάποιες μελέτες του κάποιων διαφόρων ιδρυμάτων και μιλούν για αυτά τα ατυχήματα και από το 90 μέχρι το 7 μίλταν για 2.700 περιστατικά σοβαρά που έχουν σχέση με αυτές τις υπεράκτες ε, εξορρυκτικές εργασίες και επομένως μπορεί να έχουμε σορευτικές συνέπειες των ε, μικρών επεισοδίων αλλά σορευτικά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε ε, την περίοδο εκείνη έκχυση στην, ε, και διαρροή στην Μεσόγειο 700.000 τόνων. Επομένως θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το νομοθέτημα αυτό, η οδηγία 30 του 2013. Ε, και επίσης θα πρέπει και την οδηγία 35 του 2004 να λάβουμε υπόψη που μιλά για τις ευθύνες όποτε έχουμε βλαπτικές συνέπειες προς το περιβάλλον, προς ε, χλωρίδα και πανίδα, οπότε θα πρέπει να έχουν την ευθύνη ε, οι εταιρείε ε, γιατί θα πρέπει να περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειες των εργασιών αυτών. Οπότε για αυτές τις πράκτες εργασίας χρειάζεται τελικά εξειδικευμένη νομοθεσία από τα κράτη-μέλη και να υπάρχουν επίσης έλεγχοι ενδελεχείς για να συγκρατηθούν οι συνέπειες επί προσώπων και επί του περιβάλλοντος. Συμφωνούμε με τον εισηγητή που λέει ότι δυστυχώς οι ευθύνε για ε, την πρόκληση ζημιών διαφέρει από χώρα σε χώρα. Άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις οδηγίες που ανέφερα και την οδηγία 99 του 2008 που αφορά τις ποινικέ ευθύνε ε, όταν έχουμε πρόκληση ζημιών από δόλο ή από βαρύ αμέλεια. Και να μην έχουμε επομένω ε, ρύθμιση μόνο αστική ευθύνη. Έχει δίκιο και για το νορβηγικό μοντέλο ο εισηγητέ ε, στο θέμα των αποζημιώσεων. Οπότε πιστεύω ότι με τις ε, τροπολογίες μας, στα σημεία που σας ενέφερα, ε, θα μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε το κείμενο. Γιώργος Σκοέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you. My, my name is Ευχαριστώ. Ονομάζομαι Γιώργο Κολλή. Εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πω ότι στην έκθεση που σας ε, υποβάλαμε αξιολογήσαμε την νομοθεσία η οποία ήδη υφίσταται σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση ζητημάτων ευθύνη, αποζημίωση ε, και ασφαλεία σε ό,τι αφορά τι υπεράκτε δραστηριότητε και την εφαρμογή ποινικού δικαίου ποινικών διατάξεων, όπω ήδη αναφέρθηκε. Η Επιτροπή δεν διαπίστωσε ε, κάποια γεγονότα με βάση τα οποία τα η επιβολή τη ποινική ευθύνη να μην εφαρμόζεται σε επαρκή βαθμό στα κράτη-μέλη ε, πέραν τη αστική ευθύνη. Ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα τη αποζημίωση, το οποίο αποτελεί ε, μια πολύ σημαντική πτυχή, όπω είδαμε και στι παρεμβάσει που ακούσαμε, ε, εάν θέλουμε να έχουμε περισσότερες νομοθετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να επιτύχουμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της κατάλληλης αποζημίωσης των θυμάτων και από την άλλη πλευρά ε, της ε, καταπολέμησης αξιώσεων οι οποίες δεν είναι θεμητές, δεν είναι νόμιμες. Και θα πρέπει εδώ να υπάρξει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο. Υπάρχουν δηλαδή στα κράτη-μέλη διαφορετικές παραδόσεις σε ό,τι αφορά την διάκριση μεταξύ νομίμων αξιώσεων και άλλων αξιώσεων οι οποίες ε, αποτελούν απλά απόρρια της, ε, των οικονομικών διακυμάνσεων. Αν δούμε την ίδια ε, την οδηγία και συγκεκριμένα το άρθρο 43 θα δούμε ότι τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να εφαρμόσουν διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν την άμεση και αποτελεσματική διεκπαιρέωση των αξιώσεων αποζημίωση. Εμεί λοιπόν αυτή την περίοδο από τη πλευρά τη Επιτροπή αξιολογούμε κατά πόσο τα κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει αρκούντω τη συγκεκριμένη διάταξη τη οδηγία. Για μία σειρά από σημαντικά ζητήματα υπάρχει ήδη ε, το κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά διασυνοριακού χαρακτήρα ατυχήματα. Για τέτοιου είδου ε, ατυχήματα αποφασίζεται ποια είναι η επικράτεια ε, που είναι αρμόδια για την διεκπαιρέωση των αξιώσεων ε, αποζημίωσης. Ο κανονισμός Βρυξελών 1 αναφέρει ότι ε, τα θύματα έχουν σε αυτή την περίπτωση να κινηθούν νομικά ενάντια των υπευθύνων στην αντίστοιχη επικράτεια. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται από άλλες αρχές της αλλοδαπής και με βάση τον κανονισμό Βρυξελών 2 αποφασίζεται το ποια θα είναι ε, ποιο νομικό σύστημα, ποιο νομικό, νομικό ε, το θέμα μπορεί να επιλέξει. Μετά, σε ό,τι αφορά το επίπεδο της αδειοδότηση, η Οδηγία για τα Ζητήματα Ασφαλείας προβλέπει διατάξεις σε ό,τι αφορά ε, την, ε, τι οικονομικέ δυνατότητε των ετούντων άδεια. Δηλαδή, όταν χορηγούν μία άδεια τα, οι αρμόδιες αρχέ των κρατών μελών, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, τις χρηματοοικονομικές δηλαδή δυνατότητες ε, των ετούντων για την άσκηση των ελόγων δραστηριοτήτων. Άρα λοιπόν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δεν εξετάζουν μόνο τις τεχνικές δυνατότητες ε, των ετούντων άδειες, αλλά επαληθεύουν ότι διαθέτουν τις κατάλληλες οικονομικές χρηματοδοτικές ε, δυνατότητες στο πλαίσιο αυτής της έντησης άδεια. Επίσης προβλέπεται ότι τα κράτη-μέλη και πάλι δηλαδή προβλέπεται στην ε, οδηγία εδώ για την υπεράκτη ασφάλεια, κατά πόσο ετούντα έχει ε, τις, ε, τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα για την αντιμετώπιση έκτακτων περιπτώσεων και του mediation. Επίσης, θεωρούμε πως τα κράτη-μέλη στα οποία έχουμε εκτεταμένες ε, παράκτες δραστηριότητε και άλλες ε, παράκτες δραστηριότητε, όπως δηλαδή ο παράκτος ε, τουρισμός και αλληλεία θα πρέπει να λάβουν ιδιαίτερη προσοχή. Δηλαδή θα πρέπει αυτά τα κράτη-μέλη να εξετάσουν στο πλαίσιο της ιδιαίτερης περίστασή τους κατά πόσο χρειάζεται περισσότερη νομοθεσία, πιο λεπτομερής νομοθεσία και κατά πόσο είναι θεμητή και πράγματι συμφωνώ και εγώ ότι τα όσα έχει κάνει σε αυτό το επίπεδο η Νορβηγία αποτελούν ένα πολύ καλό παράδειγμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οδηγία για το περιβαλλοντικό έγκλημα που μόλις τώρα αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις, να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε πως θα πρέπει ε, να δει ποιο είναι ο αντίκτυπο τη εφαρμογή τη οδηγία για το περιβαλλοντικό έγκλημα, με βάση δηλαδή την εφαρμογή των αντίστοιχων εθνικών διατάξεων, προτού ε, η Επιτροπή προτείνει νέε νομοθετικέ ε, πρωτοβουλίε. Τέλο, όπω προβλέπεται και στην ίδια την οδηγία, το αργότερο στο 2019 η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις εμπειρίες με βάση την εφαρμογή της οδηγίας για το περιβαλλοντικό έγκλημα και με βάση τις γνωμοδοτήσεις των εθνικών αρχών η έκθεση της Επιτροπής ενδέχεται να περιλαμβάνει τις κατάλληλες προτάσεις τροποποίησης της αφισάμενης οδηγίας και προτάσεις για την υιοθέτηση ε, περαιτέρω πρωτοβουλειών. Τα ζητήματα τα οποία θα εξεταστούν σε αυτή την έκθεση θα περιλαμβάνουν προφαλώς και ζητήματα ανάληψης ευθύνης, ε, αποζημιώσεων και ε, χρηματοδοτικής ασφάλειας προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν ελλείψεις που υπάρχουν στην εφιστάμενη οδηγία και στο πλαίσιο της επαλήθευσης της εφαρμογής της νομοθεσίας ε, η Επιτροπή θα ζητήσει από τα κράτη-μέλη ε, να ε, τις κοινοποιήσουν ποια ήταν η δική τους εμπειρία σε ό,τι αφορά τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, την αποζημίωση αλλά και τις ποινικές κυρώσεις στο πλαίσιο τη σχετική ομάδα η οποία έχει συσταθεί και η οποία συνεδριάζει τρεις φορές το χρόνο συζητώντα ακριβώ αυτό το ζήτημα τη επιβολής ποινικών κυρώσεων. Ε, ευχαριστώ. Δίνω τώρα το λόγο στον εισηγητή για τα καταληκτικά του σχόλια. Μα είναι να προλάβουμε τα όποια προβλήματα πριν προκύψουν. Η εφαρμογή του άρθρου 43 τη οδηγία δεν υποχρεώνει τα κράτη-μέλη στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Για τον λόγο αυτό και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη λήψη άμεσων μέτρων. Τώρα, η προθεσμία για τι τροπολογίε είναι μέχρι τι 3 Μαου και πιστεύω ότι μετά τη σημερινή συζήτηση έχουμε μια πολύ καλή κοινή βάση συνεργασία με όλου του συναδέλφου και του χιώδει εισηγητέ για να γίνουν τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ να υπενθυμίσω μόνο χρονοδιάγραμμα για τις τροπολογίες 3η ε, Μαΐου 12. Στην Επιτροπή ψηφίζουμε στις 11 και 12 Ιουλίου. Ευχαριστώ. Σημείο 5. Εφαρμογή νομοθεσία για την υγεία, ανταλλαγή απόψεων με του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οδηγία για τα προϊόντα του καπνού. Ξέρετε ότι η διαδικασία εφαρμογής έχει ω εξή. Ε, ε, δίνουμε το λόγο στην Επιτροπή για να αποφασίσει ε, για ποια ερωτήματα από τα 16 που έχουμε υποβάλει θα απαντήσει. Και μετά ε, δίνουμε το λόγο σε ένα από τους συντάκτες των ερωτήσεων και μετά συζητούμε. Πρώτη ομάδα ερωτήσεων ε, για τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία και την εφαρμογή. η Επιτροπή για να απαντήσει στο πρώτο ερώτημα. Ο κύριος ε, Ρή. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή. Ε, με τιμά που είμαι εδώ στο Κοινοβούλιο ε, για να συζητήσουμε την οδηγία για τα προϊόντα του καπνού που ε, στις 24 Φεβρουαρίου 2014 εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο. Ήταν ένα σημαντικό βήμα για την υιοθέτηση συνολικής προσέγγισης ε, για τα, της ε, για τα προϊόντα του καπνού για να παρασχεθεί υψηλό επίπεδο προστασίας. Φυσικά το βασικό ζήτημα είναι η εφαρμογή. Αυτό προβλέπει έγκαιρη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μεταφορά από τα κράτη-μέλη. Το 2000 ε, από το 2016 έχουν, ε, έχουν εγκριθεί πράξεις κατεξουσιοδότησης. Στην Επιτροπή για τα προϊόντα του καπνού έχουν ε, προκύψει άλλες δύο και το Μάιο περιμένουμε να γίνει το επόμενο βήμα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη παρατεταμένες περιόδους στην νομοθεσία. Ε, έχουμε ακόμη τρεις ε, περιπτώσεις ε, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου προσβάλλει την νομιμότητα της νομοθεσίας. Στις 4 Μαΐου θα εκδοθούν οι αποφάσεις την επόμενη εβδομάδα. Γερμανία για την μεταφορά στην εθνική νομοθεσία βάση των πληροφοριών που έχουμε Ε, τα κράτη-μέλη έχουν, ε, το, το Βέλγιο συγκεκριμένα, η Εσθονία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Λετωνία, η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Σλοβακία έχουν εν ή πλήρως εφαρμόσει την οδηγία από ό,τι μας έχουν ενημερώσει. Άλλα κράτη-μέλη έχουν αναφέρει ότι ακόμη μεταφέρουν τι διατάξει στην εθνική του νομοθεσία. Είναι σε διαφορετικά προχωρημένα βέβαια στάδια τη εφαρμογή συζητείται το θέμα δηλαδή ήδη στα εθνικά κοινοβούλια σε αυτές τις χώρες. Όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το ακριβές περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας ακριβώς επειδή ε, 20 Μαΐου εκπνέει η προθεσμία για τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία για να εφαρμοστεί εγκαίρωση και ομοιόμορφα αυτή η νομοθεσία από τα κράτη-μέλη. Ε, είμαστε σε διαρκή επαφή με τα κράτη-μέλη κατά τη φάση της εφαρμογής στην Πορτογαλία ε, συνεδριάζουν τακτικά οι εμπειρογνώμονες είμαστε ε, επαφή με τους ομοτήμους μας σε εθνικό επίπεδο και προσπαθούμε να καταλήξουμε συμφωνίες με τα κράτη-μέλη για τα επιμέρους σημεία. Δεν έχουμε συγκεκριμένο πρόβλημα στη Γερμανία το παρόν, αλλά μόλις γίνει ο έλεγχος, όπως σας είπα μέσα Μαΐου, θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε, λέει ο κύριος Λαβία. Ο κύριος Παγνίου μήπως θέλει να κάνει περώτηση. Ναι, Πρόεδρε. Θέλω να επανέλθω στο ρόλο της ε, του καπνού και την παρελκυστική πολιτική για τη μεταφορά τη εθνική νομοθεσία ε, προεδρεύω σε μια ειδική επιτροπή εδώ στο Κοινοβούλιο κατά της παρέμβασης της βιομηχανίας. Ε, και εξετάζουμε τις καταστρεφτικές επιπτώσεις ε, της δράσης της βιομηχανίας ακόμη και μετά την έγκριση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο του 2013 σχετικής νομοθεσίας. Χαιρετίζω τη Λίντα Μακέβεν που είναι μαζί μας σήμερα το πρωί, την ευχαριστούμε. Πήγα από το Βερολίνο στη Μεδρίτη, περνώντας από τη Βιέννη, από το Λονδίνο, από τη Ρώμη, το Παρίσι, τη Λισαβόνα, έκανα το γύρο των πρωτεύουσων και μίλησα με εκπροσώπους διαφόρων ΜΚΟ, και ε, υπονομεύει η βιομηχανία του καπνού τις ε, μεγαλεπίβολες φιλοδοξίες μας ε, πως εκφράστηκαν μέσα από αυτή την οδηγία ολόκληρη αρμάδα από λομπίστες έχουν κινητοποιήσει και έχουν γίνει σχεδόν συνομοθέτης στη διαδικασία της διαβούλευσης και οι τρεις προσφυγές που έγιναν στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της οδηγίας για το καπνό είναι το, το έσχατο παράδειγμα αυτής της ε, υποσκαπτικής ε, δράσης. Ε, Φίλιπ Μόρις και Japan, Japan Tobacco που αμφισβητούν την οδηγία προτάσσοντας ως λόγο την μη τήρηση της αρχής επικουρικότητας. Αυτή η προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της εφαρμογής της μεταφοράς στην Εθνική Νομοθεσία σε πολλά κράτη-μέλη, διότι εκεί που υπήρχε μεγαλύτερη αντίσταση σε αυτά τα κράτη-μέλη ε, χρησιμοποιούνται αυτό ως πρόσχημα για να μην ε, δράσουν. Ε, και στις 4 Μαΐου αναμένεται η έκδοση απόφασης του ΔΕ μετά ε, την απόφαση της Γενικού Εισαγγελίας της κυρίας Κοκότ ε, του Δεκεμβρίου 2015 γιατί ε, προβλέπεται ούτως ή άλλως ότι δεν ε, υπάρχει καμία παραβίαση των αρχών της αλογικότητας, της επικουρικότητας, του κράτους δικαίου και ούτω καθεξής. Οπότε θα πρέπει να επαναλάβουμε τη βούληση που μας διακατέχει να προωθήσουμε την μεταφορά στην Εθνική Νομοθεσία και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο ε, στα πλαίσια ενός δημοσίου διαλόγου και μέσω της Επιτροπής που εκπροσωπείται σήμερα να μπορέσουμε να πούμε ότι ε, ανοιχτά ότι έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα και η καταληκτική αυτή προθεσμία της 20 Μαΐου δείχνει ότι είναι σοβαρά αυτά τα προβλήματα και με τον έλεγχο της εφαρμογής θα δείτε ότι πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν συμμορφωθεί. Ευχαριστούμε. Τώρα επιπρόσθετο ερώτημα για αυτό το ζήτημα από τους συναδέλφους. Η κυρία Γκοστέτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα όλα θέλω να ξαναναφερθώ στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, διότι τελούμε να αναμονή τη έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε ε, επίση για το θέμα τη. Μισό λεπτό, μισό λεπτό διακόπτει ο Πρόεδρο ερώτηση, ερώτηση το πάμε. Οπότε υπάρχει σημείο που αφορά το λιγνωρό τσιγάρο μετά. Κύριε Γκροστέτ, ε, ξαναθέλει το λόγο. Ναι, ναι, συμπαθάτε με. Απλώς ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπε ο συνάδελφος Παρνιό για την οδηγία που αφορά τα προϊόντα καπνού. Είχαμε κάποιο διαγωνισμό και πήγε και η Οπότε, ακριβώς όπως είπε ο κύριος ε, Παρνιό, έπρεπε να ε, δούμε τις ε, συμφωνίες με τις καπνοβιομηχανίες για την απομίμηση των προϊόντων. Και ακριβώς όπως είπε η Επιτροπή, θα πρέπει αυτά τα οποία ζήτησε το Κοινοβούλιο να τα υλοποιήσει. Ευχαριστούμε ο κύριος Ντόρμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι και θέμα των λόμπι. Και είναι θέμα του κατά πόσον τηρούνται τα υπεσχημένα. Είπαμε ότι είναι υψηλή προτεραιότητα το ζήτημα αλλά τα κράτη-μέλη δεν έκαναν τα όσα ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εφαρμογή. Άρα, τι θέλει να πετύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια που δεν υπάρχει σαφήνεια στις προτάσεις της. Τι γίνεται με αυτές τις ηλεκτρονικές προειδοποιήσεις, τι θα κάνουν τα κράτη-μέλη και πώς θα το διαχειριστεί το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί επικρατεί σύγχυση. Γι' αυτό δεν έχουμε μπορέσει να τηρήσουμε τα όσα συμφωνήθηκαν εδώ στο Κοινοβουλίο. Μην ξέρω πόσο λογικό είναι οι εταιρείε να φέρουν όλες αυτές τις επιπλέον δαπάνες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ίδιο πρέπει να ισχύσει για τα αλκοολούχα ποτά, μια που επομένω τα λόμπι δεν λείπουν σε κάθε τομέα. Άρα θα πρέπει να τραβήξουμε τη γραμμή ε, ε, στο τι ζητούν τα λόμπι και τι ζητεί το κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, λέει η κυρία Ντορνάνο, όσον αφορά το διασυνορικό ζήτημα και όσον αφορά την ερμηνεία του κειμένου, θα πρέπει να περιμένουμε γιατί μα υπάρχει το θέμα στα εμπορικά ζητήματα. Είναι στην ε, τρίτη ομάδα ερωταπαντήσεων. Να το συζητήσουμε αργότερα. Να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσετε αυτές τις επιπλέον ερωτήσεις. Όπως ήδη εξηγήσαμε, έχουμε συνεχή επαφή με τα κράτη-μέλη. Τα εθνικά δίκαια έχουν επισημάνει αυτές τις προκλήσεις. Και κάποια κράτη-μέλη διάλεξαν συσκευασία απλή, χωρίς επισημάνσεις. Κάποια άλλα κρατημέλη αποφάσισαν επιπλέον μέτρα δυνάμει αυτής της νομοθεσίας. Και όπως πάντα υπάρχουν και άλλες μεταβλητές που θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι νομοθέτες. Θέματα εκτός παρασκευαστικής διαδικασίας. Εμείς πάντως θεωρούμε ότι υπάρχει βούληση για έγκριση αυτής της νομοθεσίας. Και ακόμα είναι νωρίς για να κρίνουμε ποια κράτη-μέλη θα μπορέσουν να συμμορφωθούν με αυτό το οποίο του ζητήσαμε. Εμείς πάντως είμαστε σε ετοιμότητα. States, you know, it's, uh, important to, say this is not legislation which is... Επομένως, θα πρέπει να κρατήσουμε στις αναμονές προς το παρόν, παρά ότι το πρόβλημα δεν είναι δυνατόν να χρονίσει πριν ε, θεσπιστεί νομοθεσία. Είπαμε ότι σε αυτή την περίοδο τη εφαρμογή. θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά το, το τι κάνουν τα κράτη-μέλη, όσον αφορά τις διαβουλεύσεις. Και εμείς θα προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε πάσα διαδικασία ε, και να ακούσουμε όλους τους ε, εμπλεκόμενους. Thank you very much. Uh, want to add something on Θέλετε κάτι να προσθέσετε για το δεύτερο ερώτημα που είναι η εποπτεία της εφαρμογής από τα κράτη-μέλη. Maybe I Η Επιτροπή. Ναι, όσον αφορά τα εργαλεία και μέσα πολιτικής, έχουμε τις ε, ομάδες και τις υποομάδες των ειδικών, γιατί είναι τεχνική ε, πολύ αυτή η οδηγία. Οπότε έχουμε γνωμοδοτήσεις, έχουμε διαβουλεύσεις. Όπως αυτή, αυτή την βιβλιοθήκη, το, το, το, αρχείο τέλο πάντων για αυτές τις ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις. για αυτή την επισήμανση των προειδοποίησεων. Από τρόπο δεν μπορούμε να προδικάσουμε το που θα καταλήξει αυτή η διαδρομή σε κάθε κράτος μέλος. Επίσης, αναλύσαμε τα τεχνικά μέτρα γιατί έχουμε και τους τεχνικούς ε, φραγμούς που απαγορεύονται. Και η ιστορική αγορά επιτάσσει να γίνονται κοινοποιήσεις εκ των προτέρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όποτε έχουμε έγκριση κάποιων μέτρων. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν χρειάζεται μπορεί να σχολιάσει. Ακριβώς όπως και για αυτά τα πακέτα, τη αυτή τη συσκευασία, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς επισήμανση. αιτήσει των κρατών μελών, η αιτήση δική μα. Έχουμε συνεχώ επαφέ με τα κρατημέρια. Και ακριβώ όπω είπε ε, και ο Επίτροπο. Οπότε έχουμε και αυτέ τι ε, διμερεί επαφέ που είναι πάγιο χαρακτηριστικό. Κυρία Κάντεμπαχ, θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, ένα ερώτημα στη συνέχεια των όσων είπατε. Η Επιτροπή διασφαλίζει την ύπαρξη των κατάλληλων ε, πόρων και του κατάλληλου προσωπικού για την ε, μονάδα ελέγχου των ε, προϊόντων καπνού προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά του στο επίπεδο της εποπτείας και της παρακολούθησης της εφαρμογής της νομοθεσίας της αγοράς και στο πλαίσιο της θήτη. Uh, Ευχαριστώ. Ε, κύριε Ακάλεμπα, αυτό το ερώτημα. Ναι, το ζήτημα του ανθρωπίνου δυναμικού γνωρίζετε πως αποτελεί πάντοτε ένα ζήτημα μια πρόκληση για τις υπηρεσίες της Επιτροπής καθώς βρίσκεται και μια περίοδο μεγάλων αναδιοργανώσεων. Πάντως εκείνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να προφανώς να εγγυηθούμε την συνέχεια της ομάδας για τα ζητήματα των προϊόντων καπνού και βλέπετε πως είμαστε εδώ η ομάδα με τους συναδέλφους μου για να συνεχίσουμε αυτές τις εργασίες μας. Οι προτεραιότητες μας ε, ε, προφανώς εδώ σε αυτό το τομέα αποτελούν ε, η μία από τι προτεραιότητε είναι η αποτελεσματική εφαρμογή τη σχετική νομοθεσία. Επίση συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την νομική υπηρεσία της Επιτροπής καθώς ε, και ε, με το Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο τους ώστε να υπάρχουν, υπάρχει και κατάλληλη προστασία και στο επίπεδο του δικαστηρίου της νομοθεσίας. Επίσης, θα πρέπει να, ταυτόχρονα να είμαστε προετοιμασμένοι και για τις μελλοντικέ προκλήσεις στο επίπεδο της νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι ανα πάσα στιγμή θα είμαστε σε θέση να έχουμε μια πολύ αποτελεσματική ε, ομάδα ε, σε αυτήν την ε, μονάδα και αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ καλούς συναδελφούς που συμμετέχουν σε αυτήν. Η Μπίρκετ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ένα ερώτημα έθεσα από την πλευρά μου το οποίο είναι ιδιαίτερα συναφές με αυτό το σημείο. Δηλαδή μας είπε η Επιτροπή ότι έχουμε 8 κράτη-μέλη που έχουν εφαρμόσει την νομοθεσία, τα άλλα όμως ε, ε, προχωρούν ακόμα και έχουμε και μια κατεξουσιατότηση πράξη η οποία έχει καθυστερήσει και, με βάση, ε, και στην οποία θα πρέπει να προσανατολιστεί και η εθνική εφαρμογή της νομοθεσίας αλλά όλα αυτά δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οπότε στις 20 Μαΐου θα είναι πλέον ισχύει η νομοθεσία η εν λόγω οδηγία με βάση την εθνική νομοθεσία δηλαδή πώς θα προσαρμοστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εγώ στη δικιά μου εκλογική επικράτεια έχω κάποιες επιχειρήσεις από το τομέα του τσιγαρού χαρτού οι οποίε δεν ξέρουν τι ακριβώς θα κάνουν μόλις θα τεθεί σε εφαρμογή γίνει αυτή η νομοθεσία. Ευχαριστώ. Thank you very much. Commission. Ευχαριστούμε η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Όπως είπα σε ό,τι αφορά τις διάφορες πράξεις είπαμε ότι θέλουμε να τι εφαρμόσουμε το ταχύτερο δυνατό. Για παράδειγμα σε ό,τι αφορά ε, την σήμαση και την ε, συσκευασία ή τα τεχνικά πρότυπα ε, ε, έχουν υιοθετηθεί ήδη, αλλά αυτές, αλλά ξεκινώντας από την εφαρμοστική πράξη για την ετικετοθεσία και την ε, ε, συσκευασία είχαμε μία σειρά από διατάξει που θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας και είχαμε ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2015 και ήδη από τον Ιανουάριο είχαμε δημοσιεύσει το ημερολόγιο, το χρονοδιάγραμμα δηλαδή των εργασιών μα σε σχέση με αυτέ τι πράξεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις ε, ήμασταν συνεπείς με τις προθεσμίες μας Και βέβαια στο πλαίσιο όλων αυτών των διαδικασιών χρειαζόμαστε να λάβουμε τι ε, γνώμε όλων των εμπλεκόμενων φορέων που βλέπουμε σε διαβουλεύσει με όλου του ε, stakeholders, οπότε έχουμε πάντοτε επαφέ με του εμπλεκόμενου φορέ για να ξέρουμε πότε και πώ μπορούμε να εφαρμόσουμε τέτοιου είδου ε, πράξεις. Οπότε αξιοποιούμε δηλαδή τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας για να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και η τελευταία πράξη που εκρεμεί θα έρθει σε μερικές μέρες, οπότε ελπίζω πραγματικά πως όλες, όλα τα όσα είχαμε εμείς δεσμευτεί να κάνουμε ω το Μάιο ως Επιτροπή θα έχουν λάβει χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη δέσμη ερωτήσεων. Ερωτήσεις 3 και 4, 3 και 4 που έχουν τεθεί από τον κύριο ε, Καταθούμε τα δούμε λοιπόν από κοινό αυτά τα δύο ερωτήματα και δίνω κατευθείαν το λόγο στην Επιτροπή. Ναι, έχουν να κάνουν αυτά τα ερωτήματα με την ε, εφαρμογή της ειδικής νομοθεσίας στην Ιταλία, ειδικότερα, αλλά βέβαια θέτουν ζητήματα πολύ σημαντικά για όλα τα κράτη-μέλη. Καταρχήν, όπως ήδη είπα, εμείς δεν ε, μπορούμε να σχολιάσουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας σε κάθε κράτος μέλος γιατί θα πρέπει να αναμείνουμε καταρχήν την ε, προθεσμία αυτή τη εφαρμογή στην Εθνική Νομοθεσία προτού ξεκινήσουμε την αξιολόγηση με βάση και τα όσα θα μας αναφέρουν και τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά την ανείγνευση, παρακολούθηση και ανείγνευση, το tracking and tracing, υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή, το οποίο βέβαια είναι, προβλέπει τρία ακόμα έτη, δηλαδή το Μάιο του 2019 είναι η σχετική προθεσμία. Οπότε μέχρι το Μάιο του 2019 θα πρέπει ε, οι αντίστοιχες κατεξοδότηση και εκτελεστικής πράξεις να έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή. Ε, και αυτή η περίοδος θα αποτελέσει ακριβώς το κατάλληλο παράθυρο, την κατάλληλη ευκαιρία για την υιοθέτηση των συμπληρωματικών διατάξεων στο επίπεδο της εθνικής νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη. Με βάση αυτά τα εθνικά συστήματα, αυτή η δευτερογενής νομοθεσία, νομοθεσία μπορεί να υιοθετηθεί, για παράδειγμα, μέσω διαταγμάτων των αρμοδίων υπουργών στα κράτη-μέλη. Σε συνέχεια δηλαδή των ε, συγκεκριμένων κανονισμών. Και αυτό βέβαια ισχύει ε, συγκεκριμένα για την περίπτωση τη Ιταλία, αλλά είναι πολύ πιθανό να ισχύει σε μια σειρά από περαιτέρω κράτη-μέλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα, κύριε Πεντιτσίνη, εδώ ε, μας ρωτάει κατά πόσο έχουμε λάβει πληροφορίες, δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τα νέα προϊόντα κατά τα όλα, το Product. Με βάση ε, τα όσα προβλέπει η οδηγία TPD, η εισαγωγή και η ε, παραγωγή θα πρέπει να υποβάλουν τι ειδικέ εκθέσει στι ε, αρμόδιε αρχέ των κρατών μελών και τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια μετά για τη διαβίβαση των λόγων πληροφοριών στην Επιτροπή. Αυτή είναι δηλαδή η αλυσίδα, αν θέλετε, των ευθυνών. Η Επιτροπή λοιπόν δεν έχει λάβει ακόμα αυτέ τι ε, πληροφορίε, όπω αυτέ προβλέπονται στο άρθρο 19 τη οδηγία για τα προϊόντα καπνού, τη TPD αλλά ακριβώ επειδή ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην προθεσμία τη 20η Μαου για την εφαρμογή στην Εθνική Νομοθεσία, δεν μπορούμε ε, να το αξιολογήσουμε ακόμα. Ε, δεν έχουμε δημοσιεύσει ακόμα κάποια ε, δεδομένα σε ό,τι αφορά τα νέα προϊόντα καπνού, ωστόσο τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να διαβιβάζουν τα εν λόγω, τις εν λόγω πληροφορίες, ειδικότερα σε ό,τι αφορά περαιτέρω παραμέτρους, για παράδειγμα ε, έρευνα στην αγορά, προτιμήσεις των καταναλωτών και ό,τι καθεξής. Και αυτό βέβαια αφορά όχι μόνο τα νέα, αλλά όλα τα προϊόντα καπνού και περιλαμβάνεται στις, ε, στις, στην ανάγκη της κατάλληλης προστασίας ε, της τη της ε, έτσι έχουμε σχεδιάσει το λόγο σύστημα. Σας ευχαριστούμε. Θέλετε μήπως ε, να σχολιάσετε τη παρέμβαση. Ναι, στα γρήγορα θα κάνω μία επερώτηση. Δεν θεωρώ ότι για την ε, ε ανιχνευσιμότητα μπορεί να προβλέψει τα προβλήματα που θα ανακύψουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί υπάρχουν, υπάρχει νομική πτυχή των ζητημάτων. Είναι σε εξαιρετικά δύναμη θέση οι καταναλωτές, για να, αν ε, θέλουμε να προβλέψουμε δηλαδή χρήση ενδίκων μέσων από πλευρά τους. Η Επιτροπή Ναι, ε, θα ε, εξελιχθεί το σύστημα τα επόμενα χρόνια. Λαμβάνουμε υπόψη αυτά που λέτε και θα το συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη και φυσικά με τον έλεγχο της μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία θα δούμε πώς ε, θα εφαρμοστεί ε, η ρύθμιση αυτή στην εθνική νομοθεσία και στην ε, αξιολόγηση αντικτύπου φυσικά θα γίνει διπλή επαλήθευση. αν ε, ολοκληρώσαμε για τον πρώτο γύρο να περάσουμε στο δεύτερο. Για το σημείο 5 έχουμε λάβει ήδη απάντηση. Για το 6 ενδεχομένω. Μπορείτε, ε, θέλετε να προσθέσετε κάτι ή να περάσουμε απευθείας ε, στο ερώτημα 7. Η κυρία ε, Κάτεμπαχ για την ανικανότητα μετά την κατανάλωση προϊόντων καπνού όταν κυρίως έχει αρχίσει κάποιος το κάπνισμα πριν τα 18. Αυτό είναι το ερώτημα. Πάρα πολύ σημαντικό το ερώτημα γιατί ο στόχος είναι εναρμόνιση των προϊόντων στην εσωτερική αγορά με την μέγιστη δυνατή προστασία του κοινού. Πανελειμμένα έχουμε συζητήσει το ότι η πλειοψηφία των καπνιστών ε, αρχίζουν ε, πριν από τα 18. Και τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα όσο νωρίτερα έχει ξεκινήσει κανείς το κάπνισμα. Ε, και το ζήτημα είναι τα μέτρα αποτροπής. Ε, τι έχουμε επιτύχει. Με αυτή την οδηγία έχουμε πολλά μέτρα. Παραδείγματο χάρη μεγάλες προειδοποιήσεις πάνω στα πακέτα, το κείμενο και οι φωτογραφίες που βάζουμε στα πακέτα. Είναι σημαντικό πώς διαμορφώνονται για να επηρεάζουν ε, τους νέους καταναλωτές και να τους ε, ειδοποιούν για τους κινδύνους. Προειδοποιούν για τους κινδύνους. Τα πακέτα πρέπει να είναι λιγότερο ελκυστικά. Το μέγεθος, ναι, ε, ε, όλα αυτά τα γενοτόμα ανοίγματα ή αυτά που μοιάζουν με φραγιόν, ε, όλα αυτά τα καινοτόμα πακέτα απαγορεύονται. Γιατί είναι ελκυστικά και παρακινούν τους νέους το ίδιο και για τα τσιγάρα με γεύση που στοχεύουν κυρίως το, τους νέους. Απαγορεύονται και αυτά με την νέα νομοθεσία. Μας βοηθούν διάφορα μέτρα για την προσέγγιση μας. Για τα προϊόντα καπνού που χρησιμοποιούν οι νέοι κυρίως, τα τσιγάρα και το roll your own tobacco, ο στριφτός ο καπνός, Γι' αυτό σας λέω ότι είναι στοχευμένη η νομοθεσία. Τα παρακολουθεί λοιπόν η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη πέραν αυτών και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Είναι νέο το φαινόμενο και έχουμε κατηγορίες προϊόντων που θέλουμε να μην γίνουν ελκυστικέ για τους νέους. Ενθαρρύνουμε επίσης τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τους κανόνες οδηγίες για τα προϊόντα του καπνού, ώστε να μειωθεί η πρόσβαση για τους νέους. Ε, ηλικιακό όριο, παραδείγματο χάρη, ρύθμιση ή απαγόρευση των αυτόματων μηχανημάτων ε, ε, και μέτρα που σχετίζονται με θέσεις εμπορία για αποτροπή ε, των νέων. Τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν ε, αυτό το πλαίσιο για να συζητήσουν ε, την περιπλοκότητα της κατάστασης που όπως διαμορφώνεται σε πολλά κράτη-μέλη. Ελπίζουμε να βοηθήσουμε. Και το απλό το πακέτο είναι μια νέα προσέγγιση που καθίσταται δυνατή με αυτή την οδηγία Επίσης, ε, περιβάλλον ελεύθερο καπνού, ε, ηλεκτρονικό τσιγάρο, περιορισμός της χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου στο δημόσιο χώρο, όπως ακριβώς και για τα παραδοσιακά τσιγάρα. Ευχαριστούμε. Κυρία Καντεμπάχ. Αν δεν θέλετε. Πολύ ωραία. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, επόμενη ομάδα ερωτήσεων με βατική περίοδος και καλύτερη νομοθεσία. Και πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή, όπως ήδη σας αναφέραμε, προσπαθεί να εφαρμόσει την νομοθεσια σε του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου όσον αφορά την ετικετοθεσία και τη συσκευασία με τρόπο ούτω ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί η καπνοβιομηχανία. Επίσης, τον Οκτώβριο του 2015 στείλαμε τον τεχνικό φάκελο σε όλα τα τους ώστε να ενημερωθούν. Και να υπάρξει αρκετός ε, χρόνος για τη σχεδίαση των νέων συσκευασιών σύνομα με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία. Οπότε δεν χρειάζεται, θεωρούμε, επιπλέον μεταβατική περίοδος προς την καπνοβιομηχανία. Απλώς υπενθυμίζουμε τον κύκλο ζωής του προϊόντος που είναι 6 έως 9 μήνες ανάλογα με την περίπτωση. Σχετικά ο προϊόν δηλαδή. Έχουμε την Διοργανική Συμφωνία για καλύτερη Νομοθεσία. Και οπότε θεσπίσαμε κατόπιν αυτόν την νομοθεσία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι 100% καλύφθηκαν ε, όλοι. Εμείς προσπαθήσαμε πάντως να είμαστε ανοιχτοί και να κάνουμε τη διαδικασία αυτή με διαφάνεια. Οπότε κάνουμε την ε, μελέτη των επιπτώσεων, κάνουμε τις ε, διαβουλεύσεις. Α, και τώρα για και την Παρασκευή είναι η επόμενη συνάντηση. Όπως επιτάσσει ακριβώς η Διοργανική Συμφωνία. Κυρία Γκέρλιν, δεν κάνω τη δύσκολη αλλά εδώ και 18 μήνες θέλουμε στάση αναμονής, γιατί θέλουμε να συμμορφωθούν όλα τα κρατημέλια. Αλλά, ακόμη αυτό που δεν άκουσα είναι το πώς θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα τα καταφέρει στο δεδομένο χρονοδιάγραμμα, γιατί έχουμε μέχρι τώρα πάρα πολύ λίγα κρατημέλια τα οποία έχουν ανταποκριθεί όσον αφορά την ε, μεταφορά της οδηγία, Από τον Οκτώβριο ξέρουν και έχουν λάβει τι πληροφορίε που στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχουν μεταφέρει την οδηγία στο δίκαιο του. Και δεν μιλάμε για βιομηχανία, μιλάμε για τη βιομηχανία των συσκευασιών. Στην οποία απευθυνόμεθα και λέμε ότι θα πρέπει να αναλάβει κάποιον επιχειρηματικό κίνδυνο. Αυτό δεν θα χρειαζόταν εάν γέρος είχαμε ενεργήσει. Ιδίως όσον αφορά την εξοδότηση πράξη, οι πράξεις. Αργήσαμε και είναι απογοητευτικό αυτό. Ακριβώς μια που μιλάμε για σύντομη ζωή προϊόντων. Και είπαμε ακριβώς όπως ε, επιτάσσει η οδηγία να είναι πολύ αυστηρές οι προεγραφές επισήμανσης στη συσκευασία. Είπαμε τι απαγορεύσαμε. Και τελικά θέλουμε έναν και μόνο τύπο συσκευασίας και πακέτου. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο δύσκολο να πρόκειται πιο γρήγορα. Οπότε δεν μου απαντήθηκε το ερώτημα. Μπορεί να επιβεβαιώσει η Επιτροπή ότι όλα τα κατημέλη βρίσκονται στη διαδικασία εφαρμογή. Γιατί δεν θα προλάβουμε το τέλος Μαΐου εάν δεν μπορέσουν να μεταφέρουν την οδηγία και να μπορέσουν και οι βιομηχανίες της συσκευασία να δουλέψουν επί τη βάση των όσων επιτάσσει το κείμενο του νόμου. Δεν ξέρουμε αν θα έχει γίνει μεταφορά τη νομοθεσία του ιστορικό δίκαιο. Άρα να μας πει η Επιτροπή τα κράτη-μέλη τα οποία ακόμα δεν έχουν ε, ε, ε κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις δικές τους διατάξεις θα το έχουν κάνει, θα έχουν μεταφέρει την οδηγία πλήρως ο πρόεδρος. Ο κύριος Ζόφουλ. Εκ μέρους του συναδέλφου να σας πω για το θέμα αυτό της ε, ανιγνευσιμότητας ε, των ε, καπνικών προϊόντων, όπως προβλέπετε στην εφαρμοστική πράξη της οδηγίας, διότι αναφέρθηκε για, για την προθεσμία του Μαΐου του 19 έχει γίνει μια πρώτη μελέτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη διασημότητα τον Μάρτιο του 2015 και έτσι θεσπίστηκαν ε, οι λεπτομέρειες τόσο ώστε να υπάρχει το ευρωπαϊκό σύστημα ανείχνευσης. Σήμερα δε προβλέπεται να γίνει και άλλη μελέτη. Όμως έχουμε την πρώτη μελέτη και θα πρέπει τώρα να υπάρξει το χρονικό πλαίσιο γιατί θα πρέπει να υπάρχει ανιχνευσιμότητα για να δούμε ποια προϊόντα είναι λαθρέα και τα οποία είναι επιζήμια και για την υγεία και για τους προϋπολογισμούς των κράτων μελών. Ο Πρόεδρος, αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να εξηγήσω πώς βλέπουμε εμείς ε, τις προθεσμίες αυτές και πώς μπορούν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν σωστά τις προβλεπόμενες προθεσμίες. Για τις προδιαγραφές που δώσαμε στα κράτη-μέλη τον Οκτώβριο του 2015 για όλες τις τεχνικές πληροφορίες Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να προσθέσουν αυτή την γραμμή, ε, την προειδοποιητική στο πακέτο. Με την ημερομηνία. Μέχρι την 20η Μαΐου είναι προβλέπεται η παραγωγή για να τεθεί σε εμπορία το προϊόν μετά. Πιστεύουμε ότι Ολοκληρώνουν πολλά κράτη-μέλη την ε, διαδικασία μεταφορά στην νομοθεσία και πιστεύουμε ότι εγκαίρω θα εφαρμοστεί το νέο, σύστημα. Όπως έλεγα και πριν, μπορούμε να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για τις εξελίξεις ως προς τη μεταφορά. Ε, στην νομοθεσία Όμω δύσκολα μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχο για την, ε, για την μεταφορά στην εθνική νομοθεσία. Όχι γιατί δεν επιτρέπεται, αλλά γιατί περιμένουμε και παρακολουθούμε τα προβλήματα. Και δεν γίνεται να ξεκινήσουμε πριν την 20η Μαΐου. Τώρα για την ανιχνευσιμότητα. Αρχίσαμε με τη μελέτη αντικτύπου ε, και πρέπει να περάσουμε στη μελέτη εφαρμογής. Και ε, θα κάνουμε εξωτερική ανάθεση για τη μελέτη εφαρμογής. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. όσοι θα την αναλάβουν ελπίζουμε να μας πούνε περισσότερα. Καλά, Λέω ο Πρόεδρος. Μπορούμε να περάσουμε στο τρίτο Κρούπε ερωτήσεων για τα εμπορικά ζητήματα. Μπορείτε να απαντήσετε από κοινού για τα ερωτήματα 9 και 10, γιατί σχετίζονται με το εμπόριο. Παρακαλώ. Για την ερώτηση του κυρίου Πέτερλε για την ε, σύμβαση ΠΟΕ και ε, σύμβαση που επικυρώνει είπα τώρα. Άρθρο 82 της, ε, του πρωτοκόλλου FCTC προβλέπεται όλα τα συμβολέμενα μέρη, μεταξύ των οποίων και η Ένωση, γιατί είμαστε μέλος, να έχουν ε, συστήματα ε, ανιχνευσιμότητας ε, για τα προϊόντα. Το άρθρο 812 του πρωτοκόλλου προβλέπει υποχρεώσει για τα συμβαλόμενα μέρη και για τη βιομηχανία. 16 μελούμενα μέρη έχουμε κυρώσει το πρωτόκολλο, όπω ξέρετε, μεταξύ των οποίων 5 κράτη-μέλη και η επικύρωση σε επίπεδο ένωση συζητείται τώρα στα κοινοβούλια. Αναμένεται τον επόμενο μήνα να έχουν ολοκληρωθεί οι επικυρώσει. θα γίνουν δεσμευτικέ οι διατάξει του πρωτοκόλλου για τι δράσει Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίω για την προϊόντα εργασία μα ε, για την ανιχνεσιμότητα για πράξη κατά εξουσιοδότηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας και χρειαζόμαστε τεχνικές προδιαγραφές για το μελλοντικό σύστημα αναζήτησης και ανείχνευσης. Έχουμε και τις ε, ε, ε, υποχρεώσεις του πρωτοκόλλου της μπορούμε, είμαστε σε καλό σημείο, διότι μπορούμε να συνδυάσουμε τις κατευθύντερες γραμμές του FCTC και ταυτόχρονα να εφαρμόσουμε τη δική μας νομοθεσία. Για τα ερωτήματα που σχετίζονταν με την ε, διαδικασία πέρσι, κάναμε μια στοχευμένη δημόσια διαβούλευση και αξιολόγηση αντικτύπου για το σύστημα αυτό. Δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα και Ε, σας ε, προείπα τι συμβαίνει από προς τεχνικές προδιαγραφές. Το θέμα της ε, διαφάνειας βεβαίως δημόσια διαβούλευση βάσει των σχετικών κανόνων. Ελπίζουμε να ξεκινήσει αυτό το καλοκαίρι. Και έχουμε και το εργαστήρι με όλους εμπλεκόμενους φορές. Πολύ σας ευχαριστούμε. Μήπως ο κύριος Παρνιό θέλει το λόγο. Ναι. Όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα σε αυτή τη φάση και το ότι θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση διαφήνειας και του εφαρμογή του άρθρου 100 3 όσον αφορά την σύνθεση της ομάδας των ειδικών ε, πρέπει ε, η Επιτροπή το 2017 να εγκρίνει ε, τις σχετικές κατεξοδότηση πράξεις. Ξέρουμε ότι θέλει η καπνοβιομηχανία ε, να υπάρξει και να υιοθετηθεί το δικό της σύστημα ανιχνευσιμότητας. Παρ' όλα αυτά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι είναι κατά του άρθρου 8 παραγραφός 12 του πρωτοκόλου. Που τώρα θέλουμε να νομοθετήσουμε και λέει ότι δεν θα πρέπει η καρνοβιομηχανία να παρέμβει όσον αφορά την νομοθεσία για την ανιχνευσιμότητα. Οπότε πώς θα εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η διαδικασία της έγκρισης των κατηγοριών πράξεων θα είναι όσο είναι πιο διάφανη. Γιατί έχουμε το άρθρο 123 του ΠΟΕ που ορίζει ε, τα σχετικά με την ανάμειξη των καπνοβιομηχανίων. Αυτό θα το λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κατεξοδότηση πράξεις. Thank you very much. If there are no other the floor for the Commission. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλα ερωτήματα, να δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή. Όπως σας είπα, παρακολουθούμε το πακέτο της ε, καλής νομοθέτησης Και προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατό ε, συνεπεί και να συμβουλευόμαστε τους εμπλεκόμενου, αλλά από την άλλη πλευρά είμαστε και ε, πρέπει να ακολουθούμε τα όσα ισχύουν στο κλάδο. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα ε, ζητήματα συγκρουση συμφερόντων και εμπιστευτικότητα, Οπότε, καθώς έχουμε πολλά σφαίροτα τα οποία εδώ εμπλέκονται. Από τη μία θα πρέπει να είμαστε διαφανείς, από την άλλη όμω θα πρέπει να είμαστε και αμερόληπτοι. Οπότε προσπαθούμε να επιτύχουμε αυτή την ισορροπία και είμαι βέβαιος ότι θα το συζητήσουμε αυτό το ζήτημα εκ νέου και μέσα στα επόμενα έτη. Και σίγουρα θέλουμε να είμαστε να επιτύχουμε ένα αποτέλεσμα που θα λειτουργήσει στην πράξη. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη θέση ή μάλλον στο επόμενο ερώτημα, το ερώτημα 11. Λαθρεμπόριο. Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, ε, το, η συζήτηση σε ό,τι αφορά τη συμφωνία PMI, η οποία όπως ε, γνωρίζετε έχει συζητηθεί ε, και εδώ πριν από μερικούς μήνες, είναι σχετική και βέβαια διαδέχθηκε και ένα ψήφισμα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη σχέση μεταξύ της συμφωνίας και του νομοθετικού εδώ έργου που κάνουμε, αυτό το ζήτημα συμπεριλήφθηκε και στο έγγραφο εργασίας το οποίο παρουσιάστηκε από την Αντιπρόεδρο κυρία Γεωργίευα στις 25 Φεβρουαρίου μετά από την υιοθέτηση στις 24 Φεβρουαρίου. Ε, τα όσα λοιπόν κάνει η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ σε ό,τι αφορά τις ε, διατάξεις για την ανιχνευσιμότητα ε, συνεχίζονται και προσπαθούμε στο πλαίσιο των εργασιών που κάνουμε όλα τα πακέτα των τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού να είναι ανοιχνεύσιμα ακριβώς μέσω των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας. Ε, αυτό ε, μπορώ να σας πω ε, μέχρι στιγμής, ότι δηλαδή θα προσπαθούμε να το έχουμε επιτύχει ως 20 Μαΐου του 2019. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ο κ. Πανιό θέλει να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ. Ναι. Σωστά υπενθυμίσατε ότι με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου και στα πλαίσια της σημερινή συζήτησης ε, αυτό που προσπαθούμε είναι η Επιτροπή να κάνει περαιτέρω βήματα. Μπορείτε να μας πείτε σε ποιο σημείο έχετε φτάσει, γιατί η συμφωνία με τη Philip Morris International δεν λύγει σε ένα-δύο χρόνια. Τον Ιούλη λύγει τώρα, το 16. Είμαστε τώρα ήδη στα τέλη Απριλίου. Και έχουμε και τις τρεις συμφωνίες συνεργασίας με την καπνοβιομηχανία αιτιολογούνται γιατί έχουμε και τις άλλες συμφωνίες που λήγουν το 19. Εφόσον έχουμε τα ε, εργαλεία της οδηγίας, έχουμε και το πρωτόκολλο και πρέπει να εξασφαλίσουμε την ανεκθεσιμότητα των προϊόντων καπνού μέχρι το 2017. Πώς ε, συνάδει αυτό με τις συμφωνίες αυτές. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχουν άλλα ερωτήματα, η Επιτροπή και πάλι έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ. Ναι, νομίζω πω θα πρέπει να διευκρινίσω εδώ σε αυτή τη φάση ότι έχει λάβει υπόψη τη ε, Επιτροπή την τελική απόφαση, δηλαδή σε ό,τι αφορά την μην ε, ανανέωση της ε, συμφωνία με την Φίλιπ ε, στην International. Οπότε προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να παρακολουθούμε τι εξελίξει. Euh, ε, ξέρετε ότι στο Σώμα των Επιτρόπων ε, ε, γνωρίζετε μάλλον κάτι σε σχέση με την επόμενη συνεδρία του Σώματος των Επιτρόπων, δηλαδή έχει εγγραφεί αυτό το σημείο στη μερίσια διάταξη. Απάντηση. Δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω πότε θα συζητηθεί. Το παρακολουθούμε κι εμείς. Ωραία. Το επόμενο σημείο. Επόμενη κατηγορία ερωτήσεων για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Είναι εσωτερικό το ζήτημα. Μπορείτε να αν θέλετε ε, να σταματήσουμε εδώ και αν χρειαστεί να τα κανονίσετε, να τα βρείτε μεταξύ σας αν χρειαστεί δηλαδή να θέσουμε και άλλα ερωτήματα. Πάντηση. Ναι, γνωρίζετε πως ε, αυτό το ζήτημα μας απασχόλησε στο πλαίσιο και αυτών των ε, διατάξεων και υπήρξαν μία σειρά από νομικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε ακόμα. Και θα ξεκινήσω από αυτές ακριβώς τις νομικές προκλήσεις που αναφέρθηκαν, ε, δηλαδή τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ως φαρμακευτικά συσκευάσματα. Ε, εμείς αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε να υπάρχουν σχέδια από την πλευρά οποιοδήποτε κράτη μέλους ε, να χρειάζεται άδεια για διάθεση στην αγορά ηλεκτρονικών τσιγάρων και υπήρξε μια δικαστική απόφαση ότι μια τέτοια ενιαία εφαρμογή τέτοια διάταξη όλα τα ηλεκτρονικά ε, τσιγάρα δεν ε, θα μπορούσαν να εφαρμοστεί και εδώ αναφέρομαι σε μια απόφαση του ανώτατου ε, διοικητικού δικαστήριου της Σουηδίας. Ωστόσο, αυτά τα προϊόντα θα μπορούσαν να εμπίπτουν είτε στην, στην νομοθεσία φαρμακευτικών συσκευασμάτων είτε στην νομοθεσία για ε, ιατρικά προϊόντα, αναλόγως δηλαδή με το σύστημα. Εμείς ε, ζητήσαμε από τα ε, κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την δική τους νομοθεσία τα όσα προβλέπει το άρθρο 20 της οδηγίας για, για τα προϊόντα καπνού, τα οποία προβλέπουν συγκεκριμένα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας για τα ηλεκτρονικά προϊόντα, σε όλα τα, ε, τσιγάρα, συγγνώμη, σε όλα τα κράτη-μέλη. αφού ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο εγκριθεί ως ιατρικό προϊόν, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, και είχαμε δηλαδή τη συγκεκριμένη ε, περίπτωση του ηλεκτρονικού τσιγάρου που εγκρίθηκε από τον ΕΟΦ της, του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα όσα ενδεχομένω να συμβούν και σε άλλα κράτη-μέλη. Μετά, αναφέρθηκε κάτι σε σχέση με την έκθεση αξιολόγηση κινδύνων σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Εμεί προχωράμε αυτή την αξιολόγηση σε επίπεδο εσωτερικό της υπηρεσίας και θα περάσουμε ε, στο εγγύς μέλλον στην ε, επίσημη οθέτηση μέσα στις επόμενες ημέρες δηλαδή αναμένουμε και βέβαια μόλις θα είναι έτοιμη αυτή η έκθεση θα την αποστείλουμε στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Αυτή λοιπόν η έκθεση εξετάζει ειδικότερα τους κινδύνους που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό τσιγάρο και εδώ βασιστήκαμε σε μια σειρά από πηγές πληροφοριών για παράδειγμα ε, εξωτερικούς εταίρους, ε, πληροφορίες από τα κράτη-μέλη και εμπειρογνώμονες από την ίδια την Επιτροπή. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία αυτής ε, της έκθεσης την οποία βέβαια θα λάβετε στο σύνολό τους. Καταρχήν, ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Ο πρώτος κίνδυνος είναι η κατάποση των ειδικών υγρών που περιλαμβάνουν το συλλογικό τσιγάρο και αυτό βέβαια είναι ιδιαίτερο κίνδυνος για τα παιδιά. Ε, μπορεί να υπάρξει δηλαδή ανεθισμός δερματικός ε, ε, ε, ε, ερεθισμός. επίσης υπάρχει αυξημένος πάλι κίνδυνος υγείας σε ό,τι αφορά την ανάμειξη των υγρών των ηλεκτρονικών τσιγάρων από τους, τους, τους καπνιστές και είτε ο συνδυασμός του εξοπλισμού για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είτε η συναρμολόγηση αν θέλετε ε, ε, ειδικών αν θέλετε συσκευών ε, από τους καπνιστές. Τώρα το επόμενο σημαντικό ζήτημα σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο στην υγεία και την σχετική αξιολόγηση, δηλαδή το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Πανιό, δηλαδή το πώς αξιολογούμε τον αντίκτυπο στην υγεία. Εξετάζουμε λοιπόν τον αντίκτυπο στην υγεία των ηλεκτρονικών τσιγάρων χωρίς να υπάρχει επίσημη υποχρέωση γιατί αυτή η υποχρέωση θα καλυφθεί στη σχετική έκθεση με την πλήρη έκθεση δηλαδή σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο στην υγεία των ηλεκτρονικών ε, τσιγάρων με βάση ε, τα όσα προβλέπει και η οδηγία το 2021 αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς παρόλα αυτά εξακολουθούμε να προσπαθούμε να εντοπίσουμε ε, τα νέα αναδυόμενα δηλαδή προϊόντα για των οποίων οι επιπτώσεις στην υγεία ε, δεν είναι γνωστές. Ε, συνεργαζόμαστε λοιπόν με τους αρμόδιους φορείς και εξετάζουμε προσεκτικά ε, τις πληροφορίες ε, που ε, λαμβάνουμε με βάση τις υποχρεώσεις που έχουν τα κράτη-μέλη βάσει το άρθρο 22 της TPD. Επίσης υπάρχει ένας εξωτερικός συνεργάτης ο οποίος είναι αρμόδιος για τη συγκέντρωση όλης της επιστημονικής βιβλιογραφίας σε ό,τι αφορά την χρήση των ηλεκτρονικών σιγάρων και μέσα στο καλοκαίρι θα υπάρξει και αντίστοιχη έκθεση με βάση αυτά τα στοιχεία. Επίσης, ε, το ε, νέο ε, project στο πλαίσιο του Horizon 2020 περιλαμβάνει και το ζήτημα των ηλεκτρονικών τσιγάρων και του αντικτύπου τους στην υγεία. Τέλος, σε ό,τι αφορά το ερώτημα σε σχέση με τον, τα health effects, δηλαδή τον, επιπτώσει στην υγεία, από το μέλος τεμάκι να πούμε ότι όταν ε, ε, εφαρμόσαμε για πρώτη φορά τις ε, ειδικέ υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά την ετικετοθεσία και την και τις υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά την αναφορά πληροφοριών ε, στη συσκευασία είχαμε προβλέψει ακριβώς ε, ε, τέτοιου είδους ζητήματα και περιλαμβάνουμε και στην οδηγία TPD της, την υποχρέωση να μας παρέχουν πληροφορίες ως προς το κατά πόσο το ηλεκτρονικό τσιγάρο αποτελεί μια αναλλακτική, έναν τρόπο εξοικείωση, αν θέλετε, των νέων, ειδικότερα ε, με το συμβατικό τσιγάρο. Ε, εμείς ανησυχούμε ε, σε ό,τι αφορά τον πειραματισμό των νέων με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και βλέπουμε ότι υπάρχουν μία σειρά από κράτη-μέλη τα οποία ε, θεσπίζουν ε, όρια ηλικία για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, ε, προσπαθώντα να λάβουν περισσότερε πληροφορίε για αυτά τα προϊόντα. Όμω ταυτόχρονα βλέπουμε και πολύ ανησυχητικέ τάσει, για παράδειγμα από τι ΗΠΑ, όπου από το 2011 έω το 2015, δηλαδή μόνο σε περίοδο 4 ετών, μεταξύ των ε, μαθητών ε, του Λυκείου το ποσοστό των καπνιστών ηλεκτρονικών τσιγάρων αυξήθηκε από 1,5% σε 16% και από 0,6% σε 5,3% αυξήθηκε το ποσοστό των, ε, των καπνιστών ηλεκτρονικού τσιγάρου στα γυμνάσια. Αυτά είναι βέβαια, όπως σας είπα, δεδομένα τα οποία έχουμε λάβει από τις ΗΠΑ Τώρα, γιατί δεν υπάρχει κάποια μελέτη αντίστοιχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σας είπα πάντως πως τα πορίσματα της σχετικής έκθεσης ε, θα είναι σύντομα διαθέσιμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, την ε, προστασία των μη καπνιστών και την έκθεσή τους, δηλαδή στον καπνό των καπνιστών, να πούμε ότι η νομοθεσία που αφορά τα περιβάλλοντα απαλλαγμένα από καπνό αποτελεί ε, ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας. Οπότε εμείς καλούμε από τα ε, κράτη-μέλη να ε, λάβουν αντίστοιχες, αντίστοιχες, να προβούν σε αντίστοιχες διατάξεις, αντίστοιχη νομοθεσία. Υπάρχουν ερωτήματα. Ζήλ. Ε, τίποτα να ευχαριστήσω θέλω για τις απαντήσεις σας, διότι βλέπω ότι παρακολουθείτε από πολύ κοντά και μελετάτε τις ε, μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου. η έκθεση, από ό,τι κατάλαβα, που έπρεπε να έχει διαβαστεί στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μέχρι τις 20 Μαΐου, θα δημοσιευθεί ε, το καλοκαίρι. Ελπίζουμε το ελπίζουμε, διότι το είπανε και οι συνάδελφοι, είναι πρόβλημα ε, δημόσιας υγείας, κυρίως, ναι. κυρίως ε, για τους νέους. Ε, διότι υπάρχει το πρόβλημα της ε, δυνάμει χρήση ε, των καταναλωτών από τους νέου και εφόσον δεν θεωρείται προϊόντο ε, προϊόν που μας βοηθάει να κόψουμε το κάπνισμα, ένα ε, φαρμακευτικό σκεύασμα, όπως είπε εξάλλου και η καπνοβιομηχανία, <clears throat> θέλει να συμμετάσχει στη διαβούλευση για την πώληση των τσιγάρων, ώστε ε, να μπορέσει να επηρεάσει τα υγρά που το μείγμα των υγρών μέσα στο ηλεκτρονικό τσιγάρο ε, γιατί δημιουργείται θυσμός στους νέους, ε, ισχυρότατος θυσμός με την νοικοτήνη. Ξέρετε ότι την προηγούμενη θητεία εμείς ζητήσαμε να θεωρηθεί σκεύασμα σχεδόν φαρμακευτικό που χρησιμοποιείται στο τομέα της υγείας το ηλεκτρονικό τσιγάρο και ελπίζοντας ε, έτσι να ισχύσουν αυστηρότεροι περιορισμοί για την πώληση ε, των προϊόντων αυτών, επειδή θεωρούνται ως ε, φαρμακευτικό σκεύασμα, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστούμε, κυρία Γκροστέ. Ναι, Όπως είπε και ο κύριος ε, Παρνιό, όταν ε, διαπραγματευόμασταν αυτή την οδηγία, ξέραμε πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να πιέσουμε πολύ για την νομοθεσία και δεν υπήρχε μεγάλο περιθώριο βελτίωση διότι υπήρχε θέμα εναρμόνιση. Εάν μας λέτε ότι είναι σοβαρός ο κίνδυνος για την υγεία, τότε θα πρέπει όλοι να ε, δεχτούμε να τοποθετηθούμε για το ηλεκτρονικό τσιγάρο και να ε, έχουμε μια διαφορετική εναρμονισμένη ρύθμιση σε επίπεδο ένωσης. Ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα του εθισμού στην νοικοτήνη που προκαλείται από αυτή την ε, χρήση, από τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Όντως, το ταχύτερο δυνατόν θα θέλαμε να έχουμε αυτή την έκθεση, πάντως μόλις εκπονηθεί αμέσως θα πρέπει να ε, επιληφθούμε του ζητήματος για να δούμε τι θα κάνουμε με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος να προσθέσει οτιδήποτε σε σχέση με αυτές τις ερωτήσεις. Τότε η Επιτροπή. Τώρα Μιλούμε για τους κινδύνους από τα λιγνά τσιγάρα που θα έχουμε την έκθεση τον ε, Μάιο και θα έχουμε επομένω την επιστημονική γνωμοδότηση και έτσι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις γνώσεις μας. Λόγοντας που πονού όλη την επιστημονική ύλη. Βεβαίως θα πρέπει να γίνει κάποιο είδους μακρόπνοη ε, παρακολούθηση θέλουμε πέντε χρόνια να παρακολουθήσουμε τι γίνεται με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Όπως είπε και η Να μπορέσουμε έτσι στη συνέχεια να αναθεωρήσουμε τη σχετική νομοθεσία. Πάντως θα πρέπει και με λόγο οδηγία ε, να την ε, εφαρμόσουμε και τότε θα μπορέσουμε επίση να συλλέξουμε πολλά στοιχεία. Τότε θα είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να επανέλθουμε στο θέμα ε, στο μέλλον. Κυρία Γκροστέ, θέλετε κάτι να συμπληρώσει, ναι. Ε, μου φαίνεται όμω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο χρόνο διάστημα η πενταετία, γιατί τότε είναι θέμα υγεία. Δεν επιτρέπεται τόσο πολύ να περιμένουμε. Οπότε ελπίζω ότι μπορούμε να πιέσουμε ούτω ώστε το θέμα αυτό να διεκπαιριωθεί και να προχωρήσει ταχύτερα. Μόλις ε, ολοκληρωθεί η έκθεση να μπορέσουμε συντομότερα να τα δούμε και να μην περιμένουμε όπως πάντα εκθέσεις επί εκθέσεων και εξέταση αυτών κλπ. Είναι θέμα υγείας, δεν περιμένει. Thank you very much, Ms. I don't know if the commission... Ευχαριστούμε κύριε Δεν ξέρω Θέλει κάτι να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Καλώς. Πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα. Αφορά, τελευταία ερώτηση, το περιεχόμενο. Έχει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ερώτηση του κυρίου Φλόρεντς. Πώ ερμηνεύουμε το άρθρο 7, παραγράφο 7. Πρώτα πρώτα. Αυτά τα στοιχεία είναι η εσωτερική αξιολόγηση της Γενικής ε, Διεύθυνσης για την ε, Υγεία. Δεν δεσμεύει την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε είναι αυθεντική ερμηνεία της οδηγίας που γίνεται μόνο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πάντως, σύμφωνα με τη δική μας ερμηνεία, τέλο πάντων την ερμηνεία της Διεύθυνσης για την Υγεία, αυτά τα οποία ορίζει το άρθρο 7 παραγράφος 4 σημαίνουν ότι η οδηγία δεν ισχύει για αυτά τα μέρους περιχώμενα όπως φίλτρα και πρόσθετα αρωματικά και γευστικά. Οπότε έχουμε τη σχετική παρέκκληση και λέει για κάποια προϊόντα τα οποία θα καταργηθούν βαθμία ούτως ώστε να μπορέσουν οι καταναλωτές να κατευθυνθούν προς άλλα προϊόντα. Και όταν κάποια προϊόντα έχουν ικανό μερίδιο αγοράς, έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση, μεγαλύτερο δηλαδή διάστημα της ε, σταδιακής κατάρριξης για να πάνε αλλού οι καταναλωτές. Ο δε στόχος να έχει αρκετό χρόνο ο καταναλωτής για πέσει άλλο προϊόν λέει ότι δεν δικαιολογεί άλλη ρύθμιση για τα φίλτρα κλπ και ένας από τους στόχους της είναι η πρόληψη της εξάρτησης από το κάπνισμα για τους νέους και αυτές οι καψούλες είναι ελκυστικές και επομένως ελκύουν κατάλληλοι ότι αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω ο κύριος ε, Φλόρενς ε, θέλει να απαντήσει κάποιο άλλο, άλλο συνάδελφος. Εάν όχι, νομίζω πως ε, μπορούμε να κλείσουμε με τη συνεδρίαση της Επιτροπή μας. Να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσία της εδώ και τις απαντήσεις που μας έδωσε και τις διευκρινήσεις που λάβαμε. Σήμερα το απόγευμα στις 3 ε, ε, η ώρα θα συνεχίσουμε με το δεύτερο τμήμα της συνεδρίασής μας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους.